Good afternoon. welcome to the... Καλώς ορίσατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Κανονικά πρέπει να αρχίσουμε από το 15, αλλά ε, έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση και στους συντονιστές και στους υπολείπους συναδέλφους της Επιτροπής μας σχετικά με τη γραπτή διαδικασία για τις νέες μελέτες που θα αναθέτουμε από την Επιτροπή μας. Έχουν εγκριθεί τα εξής θέματα από τις πολιτικές ομάδες. Πρώτον, μελέτη για την ενημέρωση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενημέρωση της μελέτης του 2004. Δεύτερον, μελέτη για το μέλλον της Eurojust. Τρίτον, σημείωμα για την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την καταπολέμηση αυτή. Τέταρτον, σημείωμα για την ανάγκη για νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να επιτρέπει τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί γιατί είναι προϊόντα εγκλήματος να μπορούν να χρησιμοποιούνται από την κοινωνία των πολιτών για κοινωνικούς σκοπούς. Στη συνέχεια, σημείωμα για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτο ήταν αυτό. Έκτο, σημείωμα για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, για κάποιους οργανισμούς ε, Frontex, Europol, ορισμένες πολιτικές ομάδες ζήτησαν να ξανακοιτάξουμε μία από τις μελέτες που είχαμε προτείνει, αν είναι σκόπιμη, και ή να προτείνουμε νέες ιδέες. Θα τα επεξεργαστούμε όλα αυτά και θα επανέλθουμε στους συντονιστές με νέες προτάσεις το συντομότερο. Αυτά. Όχι, δεν είναι αυτά. Έχουμε κι άλλα. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στο σημείο 15. Όχι, αλλά έχουμε πρώτα το 14. Θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν. Έχουμε εδώ ένα θέμα του οποίου εισηγητής ο Κάρλος Κοέγιο έχει εργαστεί πολύ χρόνο και τώρα έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων παρουσία εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σούστρο και τον κύριο Ντεμπάρ. Ε, καλώς στην Επιτροπή μας. Και όπως σας είπα, κατόπιν πρωτοβουλίας του κυρίου Κοέγιο προσκαλέσαμε τους δύο εμπειρογνώμονες και τον κύριο Σούστρο που είναι Τσέχος εκπρόσωπος ε, του Υπουργείου Ιστορικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης ε, στην υπηρεσία αξιολόγηση του Σέγγεν, στην ομάδα εργασία. Και ο κύριο Πατρίκ Ντεμπέρ είναι ο Γάλλο εκπρόσωπο στην ομάδα εργασία για την αξιολόγηση του Σέγγεν. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο πρώτα στον εισηγητή μα, μετά στου υπηρογνώμονες σύντομες παρεμβάσεις και μετά την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση ως συνήθως με τα μέλη της Επιτροπής μας. Κύριε Κοέγιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονε που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και ήρθαν στη συνεδρίαση αυτή. Θέλουμε ένα μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν που θα βελτιώνει το υπάρχον σύστημα, θα το απλουστεύει, θα το, θα το καθιστά αποτελεσματικότερο και ένα γνήσιο ευρωπαϊκό σύστημα. Προτείνω να ακούσουμε αμέσως τους εμπειρογνώμονές μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας εκθέσουν τα σημαντικότερα κατά τη άποψή τους θέματα και θα τους παρακαλούσα οι δυνατόν να δώσουν απαντήσεις σε τρία θέματα που είναι αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις, τις διπλές προδιαγραφές. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ένα ε, μηχανισμό αξιολόγησης ό,τι αφορά την προηγούμενη επαλήθευση, εκ των προτέρων ε, ε, επαλήθευση για τους υποψήφιους και μετά ένα μηχανισμό αξιολόγησης ε, για τους χώρες που είναι ήδη μέλη του χώρου Σέγγεν. Ερωτώ λοιπόν, δεν είναι σκόπιμο να έχουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς ε, διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ υποψήφιων χωρών και το χώρο Σέγγεν και χωρών μελών του χώρου Σέγγεν. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις συνέπειες για τις υποψήφιες χώρες ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες μιας αξιολόγησης. Αν είναι αρνητική αξιολόγηση δεν δικαιούνται να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Για τις χώρες που είναι όμως ήδη μέλη του χώρου Σέγγεν δεν ε, απορρέουν συνέπειες από μια αρνητική αξιολόγηση. Ερωτώ λοιπόν, μήπως θα πρέπει να θεσπίσουμε και κυρώσεις που να επιβάλλονται στις χώρες που είναι μέλη του χώρου Σέγγεν σε περίπτωση που το πόρισμα της αξιολόγησης είναι αρνητικό και που καταδεικνύει σοβαρές αδυναμίες ε, τέτοιες που να θέτουν ε, αναφιβόλω την ασφάλεια στο χώρο Σέγγεν. Και η τελευταία ερώτηση αφορά τις παρατηρήσεις που έκαναν ορισμένοι συνάδελφοι της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που ζήτησαν να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια στην αξιολόγηση του Σέγγεν. Για παράδειγμα, η εμπιστοσύνη στον έλεγχο που κάνει στα εξωτερικά σύνορα μία χώρα δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των ελεγκτών ε, ή από τον αριθμό των δερματικών για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια που να καθορίζουν την εμπιστοσύνη που θα έχουμε στη, στη χώρα που πραγματοποιεί τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, ώστε να αισθανόμαστε πραγματικά ασφάλεια στο χώρο του Σέγγεν. Ερώτηση λοιπόν είναι σκόπιμο να προσθέσουμε και άλλα κριτήρια και ναι πια για το νέο σύστημα αξιολόγηση του Σέγγεν. Αυτέ είναι οι ερωτήσει μου. Ευχαριστώ και προτείνω να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονέ μας. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Και τώρα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρτιν Σούστρου και θα τον παρακαλέσω να μιλήσει να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση για να ακούσουμε στη συνέχεια και το δεύτερο πυρογνώμονα και μετά να γίνει συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε όλους. Καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και τον Πρόεδρο και τον εισηγητή που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την άποψή μου για ε, την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να σας πω ότι σε κάποιο βαθμό ε, η προσωπική μου θέση ταυτίζεται με τη θέση της Τσεχικής Δημοκρατίας. Όπως γνωρίζετε είμαι εκπρόσωπος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση και πριν έρθω στα τρία θέματα και στις τρεις ερωτήσεις επιτρέψτε μου σύντομα να σας κάνω μια σκιαγράφηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της πρότασης όπως εμείς την αξιολογούμε. Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες σήμερα. Το σημαντικότερο είναι το θέμα της παρακολούθησης, η συνέχεια που δίνεται στην αξιολόγηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν σχόλια και να ε, ε, στέλνουν αναφορές για τις αλλαγές που έγιναν με βάση ε, τις συστάσεις. Σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα αντίδραση εάν δεν βελτιώνει μια χώρα μέλος την κατάστασή της κατόπιν των συστάσεών μας. Και αυτό έχει βεβαίως μεγάλη επίπτωση σε άλλα κράτη Σέγγεν. Και αν ένα κράτος ε, Σέγγεν δεν συμμορφώνεται με το κεκτημένο και τι υποχρεώσεις, αυτό έχει ε, επιπτώσει για όλα τα υπόλοιπα κράτη του Σέγγεν. Τα οποία κράτη Ε, χρειάζεται εκ των υστέρων να επιβάλλουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και άλλα τέτοια μέτρα. Και ως αποτέλεσμα αυτό αποδυναμώνει σημαντικά την ποιότητα ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που είναι ε, διανόμου συγγνώμη, κατοχυρωμένη και εγγυημένη. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κομβικά ζητήματα. Το κεντρικό θέμα του Σέγγεν είναι η έλλειψη των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες και τα παράπονα των πολιτών, έχουμε ερωτηματικά. Εάν και κατά πόσο αυτά πάντα συμβαίνουν που καταγγέλουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται εδώ να σας τονίσω τα προβλήματα, ούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, ούτε την ασφάλεια που ανήκουν ε, στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αξίες που τόσο πολύ τις εκτιμούμε και δεν θα πρέπει να διακυβεύονται. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξετάζει αυτά τα θέματα με το σωστό τρόπο και στην παρακολούθηση και στη συνέχεια που δίδουν και ε, όπως έδειξε η πρόσφατη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών μπορεί να ανοίξει συζήτηση για δυνατότητα ε, αναστολής της συμμετοχής μιας χώρας στο Σέγγεν σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων. Θα επανέλθω σε αυτό. Ως Ευρωπαίος πολίτης χαίρομαι για την αξιολόγηση που έγινε για τα εσωτερικά σύνορα, όπως ε, προτείνει το άρθρο 12. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός των εσωτερικών μας σύνορων και η διαφύλαξη αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να είναι αντικείμενο του μηχανισμού αξιολόγησης. Επειδή εκπροσωπώ και ένα κράτος μέλος, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αυτό το άρθρο μπορεί να ε, τροποποιηθεί μόνο για να συμμετέχουν και άλλοι εθνικοί πυρογνώμονε εκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε, να σα πω μόνο κάποια άλλα θετικά που άλλαξαν προς τη σωστή κατεύθυνση η ανάλυση κινδύνου που κάνει Frontex ή η ε, επιστροφή των εξόδων εμπειρογνωμόνων των ε, κρατών μελών, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η περισσότερη συνέργεια στη συνεργασία σε θέματα Σέγγεν. Επίσης, αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε και άλλα αιτήματα που είναι κοινά πολλών ε, κρατών μελών, όπως οι χώρες του Φόρουμ του Στρασβούργου και το αίτημα να διατηρηθεί η σημερινή πρακτική ε, ακριβώς ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών και με ένα μηχανισμό ε, νέο, όχι πριν το 2014 όταν θα ολοκληρωθεί το τρέχον πενταετές πρόγραμμα αναθεώρησης. Για ποιο λόγο το τρέχον πρόγραμμα ισχύει μέχρι τα τέλη του 2013 και είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνε σε όλα τα κράτη-μέλη του Σέγγεν με τον ίδιο τρόπο και το καινούριο πρόγραμμα να αρχίσει με του νέου κανόνε. Επιτρέψτε μου τώρα σύντομα να αναφερθώ σε τρία άλλα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα και θα νομίζω μας χρησιμεύσουν στον προβληματισμό μας, τα είπε και ο κύριος Κοέλιο, διαφορετικό μηχανισμό αξιολόγησης που έχουμε άλλο για τα κράτη-μέλη και άλλο για τα υποψήφια κράτη-μέλη. θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα τα κράτη-μέλη, να ελέγχουν τα υποψήφια κράτη και ε, να αξιολογούν αν και κατά πόσο ε, πληρούν τις τα προαπαιτούμενα και τις απαιτήσει για να ενταχθούν στο Σύνταγμα Σάγγεν και αυτά εκ των προτέρων να μην αλλάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γιατί έτσι μόνο εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση. Για να ε, εγγυηθούμε ότι υπάρχουν τα ίδια κριτήρια, το μέσο ειδικής αξιολόγηση του κεκτημένου Σέγγεν και των βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να διατηρηθεί. Εν πάση περιπτώσει, η συνύπαρξη δύο επιτροπών, η Επιτροπή της Επιτροπολογίας και η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου δεν είναι τίποτα νέο. Συμβαίνει και αλλού στη συνεργασία Σέγγεν, για παράδειγμα στα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων, όταν έχουμε την Ομάδα Εργασίας ε, για ε, τις θεωρήσεις και την Επιτροπή για τι θεωρήσεις. Ε, επίσης, τώρα, ε, αν στην αξιολόγηση ε, είδαμε αδυναμίες ε, στις ε, διαδικασίες, όντως, και ε, χωράει βελτίωση αυτή η διαδικασία, οι νέοι κανόνες θεωρητικά μπορούσαν να οδηγούν μέχρι και αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν ε, σε κάποια κράτη και άλλες κυρώσεις μη οικονομικού χαρακτήρα. Όσα ε, και είναι δύσκολο αυτό να υλοποιηθεί έτσι από πλευράς πρακτικής θα πρέπει να διατηρείται πάντα η αμοιβαία εμπιστοσύνη και κάθε κράτος μέλος να θεωρεί υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του. Δυστυχώς σήμερα η ε, κυρώσεις περιορίζονται σε κάποιες επισκέψεις ε, σπάνιες και παροδικές, αλλά και αυτό δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Τα κριτήρια θα πρέπει να γνωρίζουμε, απλώς θα το μιλούμε για ένα μηχανισμό που αξιολογεί το κεκτημένο του Σέγγεν. Γι' αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζεται σε μέτρα ε, του κεκτημένου του Σέγγεν και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες. Βεβαίως, στο μέλλον δεν αποκλείεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή Πάντα μέσα στα πλαίσια του κεκτημένου του Σέγγεν. Παράδειγμα, κατά πολέμηση του οργανωμένου κλίματο ή της διαφθοράς, όπως ε, σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στο Σέγγεν θα, θα το αξιολογούμε και αυτό, αλλά όχι εκ των προτέρων. Τώρα μας απασχολεί μόνο το κεκτημένο του Σέγγεν. Θα περιοριστώ λοιπόν ολοκληρώνοντας να πω ότι ε, βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο στη συζήτηση αυτή και ορισμένα άλλα στοιχεία ουσιώδη της πρότασης, όπως είναι η, λογική, η νομική βάση, συγγνώμη, η συμμετοχή του Εμμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, δουν και να αξιολογήσουν ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις διάφορες ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις και μεταξύ αυτών και στη σημερινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Monsieur Patrick Ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ντεμπέρ, τον Γάλλο εκπρόσωπο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία σε έναν Γάλλο εμπειρογνώμονα να εκφράσει την θέση της χώρας που εκπροσωπεί. Θα σας παρουσιάσω την γαλλική θέση η οποία συμπεριλαμβάνει πέντε βασικά σημεία. Και θα κάνω ένα αρχικό σχόλιο λέγοντας ότι εμείς είμαστε υπέρ αυτού του νέου μηχανισμού που προτείνει η Κομισιόν αλλά πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος για να μπορέσει δηλαδή να επιφέρει μια μεγαλύτερη, να, να περισσότερη υπεραξία στη διαδικασία Σέγγεν. Αυτό το οποίο θέλουμε σε αυτόν τον νέο μηχανισμό είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν. Και αυτό φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή εμπειρία της αξιολόγησης Σέγγεν και τα όρια της. Η Κομισιόν θα επιτρέψει μέσα από την ανάλυση των συστάσεων αλλά και από την αξιολόγηση θα μπορέσει να συνεισφέρει με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία Περισσότερο δηλαδή από ότι σήμερα τα κράτη-μέλη που επεξεργάζονται τις συστάσεις. Επίσης ενισχύεται και η αντικειμενικότητα αυτών των εκθέσεων αξιολόγησης. Αυτή είναι η πρώτη άξονα σκέψης που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε με τον νομιχανισμό. μηχανισμό. Δεύτερη επιθυμία που θέλουμε να ληφθεί υπόψη είναι να δοθεί ένας ιδιαίτερος ρόλος, ένας πιο σημαντικό ρόλος στους ε, κοινοτικούς οργανισμούς. Σε δύο φάσεις του μηχανισμού αξιολόγησης Schengen. Στην φάση δηλαδή της ε, σύνταξης, η Frontex, η Europol και η Eurojust να παίξουν ένα ρόλο υποστήριξης σε αυτήν τη διαδικασία. η Frontex να παίξει ένα ρόλο στη φάση προετοιμασίας, ε, η Europol να συνεισφέρει με την ανάλυση του ρίσκου, η Frontex ε, για παράδειγμα όσον αφορά στα μεταναστευτικά κύματα και η Europol ε, στο οργανωμένο έγκλημα και μετά να μπορούν στην επόμενη φάση να συνεισφέρουν στην ίδια την αξιολόγηση με παρατηρήσεις. Ένα τρίτο στοιχείο απαντά και σε μία από τις ερωτήσεις του Προέδρου. Σήμερα ο μηχανισμός αξιολόγησης όταν διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν δεν οδηγεί στη λήψη πραγματικών κυρώσεων. Εκτός πια και αν ασκηθεί η δυνατότητα της Κομισιόν η οποία μπορεί να ασκήσει προσφυγή παραλήψη. Αλλά στην τωρινή φάση Το μόνο που γίνεται είναι νέες επισκέψεις αξιολόγησης και δεν, δεν υπάρχει κάτι το κατασταλτικό. Όταν δηλαδή γίνονται συστάσεις μετά από την αξιολόγηση και αυτές οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα κυρώσεων για να μπορέσει να ενισχυθεί ο χαρακτήρας των αξιολογήσεων. Και οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν και μια αναλογία, μια αναλογικότητα με τις ελλείψεις που διαπιστώνουν οι αξιολογητές. Εμείς ε, στη γαλλική διοίκηση προβληματιζόμαστε γύρω από ορισμένες ε, κυρώσεις, ο συνάδελφός μου ανέφερε ορισμένες ε, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στον αποκλεισμό ενός κράτους μέλους από το Σέγγεν. Αλλά ακόμη δεν αποφασίσαμε τι είδους κυρώσεις ε, θα θέλαμε να προτείνουμε στο πλαίσιο αυτού του νέου μηχανισμού αξιολόγησης. θα συνεισφέρουμε όταν έρθει η ώρα για αυτό το θέμα. Αλλά επί της αρχής εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχει ένα σύστημα κυρώσεων, όχι μόνο ε, για τις κυρώσεις αυτές καθεαυτές, αλλά να παίζει και έναν προληπτικό ρόλο έναντι των αξιολογουμένων κρατών. Ένα άλλο σημείο, το οποίο θα επιθυμούσε η Γαλλία, είναι στο νέο μηχανισμό να έχουμε δύο καθεστώτα, αφενός δηλαδή την αξιολόγηση για τις χώρες εκείνες οι οποίες εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σέγγεν και δεν εφαρμόζεται όμως πλήρως στις χώρες εκείνες οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη του Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μία διαφορά κατηγοριών μεταξύ των χωρών εκείνων που εφαρμόζουν πλήρως ε, το κεκτημένο του Σέγγεν και αυτών που δεν το εφαρμόζουν πλήρως, γιατί αυτό δεν θα είχε νόημα. Και βασίζομαι σε αυτά που είπε ο προλαλής και ε, ότι δηλαδή υπάρχει μία ενότητα καθεστώτους, και επαλήθευσης της εφαρμογής του Σέγγεν. Γιατί αν υπάρχει αυτή η διπλή κλίμακα αξιολόγηση, οι πρώτοι θα έχουν την τάση να γίνουν δεύτεροι μετά. Και αυτό θα ζημίωνε όλο το χώρο Σέγγεν και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών το επόμενο σημείο που θα θέλαμε είναι ένα σημείο που ήδη αναφέρθηκε. Μέσα στο εφαρμοστικό πεδίο του νέου μηχανισμού να συμπεριλάβουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία τίνουν μέσα στο πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης να ευνοούν την ελεύθερη κυκλοφορία. Υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να προστατεύσουμε οπωσδήποτε και αποτελεί το θεμέλιο, τη βάση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Θα θέλαμε λοιπόν πέρα από την τωρινή αξιολόγηση Schengen, δηλαδή προστασία των δεδομένων, σύστημα πληροφόρησης, σύστημα ε, ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, αστυνομική συνεργασία, θα θέλαμε να προστεθεί και η αξιοπιστία, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας, της ε, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, όπως επίσης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Συνολικά δηλαδή όλα εκείνα τα κριτήρια τα οποία επιτρέπουν να εγγυηθούμε ότι μέσα στο χώρο Σέγγεν θα προστατεύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών Σέγγεν. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο στοιχείο για τη συνεργασία. Αυτά κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα και είμαι βέβαια και στη διάθεσή σας, όπως και στη διάθεση των βουλευτών, για να αναπτύξω περαιτέρω ορισμένα σημεία. Αυτοί είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η γαλλική διοίκηση και επιμένω ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι διότι θα πρέπει να μπορέσουμε να δυναμώσουμε, να σταθεροποιήσουμε το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην ζώνη Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντεμπέρ. Περιμένουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, αν θέλουν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Ίσως πρώτα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου την, την κυρία Τιμία Άντεξ ή δεν θέλει να λάβει το λόγο. Κανείς από, το προεδρία, από την Προεδρία. Μήπως έκανα λάθος το όνομά σας. Καλά πείτε μας πώς λέγεστε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω λίγα λόγια για το έργο που γίνεται στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο και θα γνωρίζετε ότι στα τέλη της Βελικής Προεδρίας ε, υπευλήθη πρόταση του Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής έγιναν λίγες διαπραγματεύσεις και μέχρι στιγμής ακροθυγώς έχουμε εξετάσει την πρόταση. Πάντως εκ πρώτης όψης φαίνεται τα κράτη-μέλη είναι υπέρ των προτάσεων για την ενίσχυση και τη βελτίωση του μηχανισμού αξιολόγησης. Προς το παρόν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η μέχρι τώρα εμπειρία μας θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στη νέα πρόταση. Για παράδειγμα, Λίγες χώρες μέλη είναι υπέρ της πρότασης να προσδιοριστούν οι χώρες στις οποίες θα αποστέλλονται οι εμπειρογνώμονες. Να είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση δηλαδή για το ποιο θα στέλνεται. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση τη απορρίμηση του μηχανισμού αξιολόγηση να περιληφθεί και η Frontex. Και οι περισσότερε χώρε μέλη είναι υπέρ αυτή τη πρόταση. Η Frontex, ο οργανισμός Frontex θα συμμετέχει και θα συνεργάζεται στην ανάλυση του κινδύνου και θα συμβάλλει και στην κατάρτιση του προγράμματος της ετήσιας αξιολόγησης. Επίσης διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι δράσεις θα πρέπει να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ των δράσεων των εθνικών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να ελέγχεται η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή την άποψη υπάρχει διάσταση απόψεων στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Ένα τμήμα των μελών τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου θεωρεί ότι δεν ε, έχει νόημα να γίνεται και εσωτερικό έλεγχο, ενώ άλλες χώρες στην ομάδα εργασίας πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην εξελόγηση αυτή όχι μόνο εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της επιτροπολογίας, αυτή τη διαδικασία προτείνει το Συμβούλιο για να συμπεριληφθούν και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Βέβαια, πολλές χώρες μέλη είναι αρκετά επιφυλακτικές προς την πρόταση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέα διαδικασία επιτροπολογία στην επόμενη συνεδρίαση. Φαίνεται όμως ότι τα κράτη-μέλη εν αναμονή της νέας πρότασης δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει τη γνώμη τους. Θα περιμένουν την πρόταση αυτή για να λάβουν θέση. Ελπίζω ότι θα γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση στην επόμενη συνεδρίαση γιατί βρισκόμαστε ακόμη σε πρόωρο στάδιο της διαδικασίας και τότε ελπίζω να σας ενημερώσω και πιο διεξοδικά. Θα ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μόνικα Μοσάμερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή σας και τον εισηγητή για την πρωτοβουλία. Γιατί καλό είναι που έχουμε όχι μόνο τεχνική αλλά και συζήτηση επί της ουσίας της πρότασης. Εγώ θα επικεντρωθώ στις τρεις ερωτήσεις του εισηγητού. Σε ό,τι αφορά τα διαφορε... τις διαφορετικές προδιαγραφές, τις διπλές προδιαγραφές, εμείς στο νέο μηχανισμό αξιολόγησης για, το δεύτερο τμήμα, δηλαδή για την άρση του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα, έχουμε τη νέα πρόταση. Ανάλογα με την συνθήκη προσχώρηση έχουμε διαφορετική κατάσταση και διαφορετικές απόψεις όπως φάνηκε από τους εμπειρογνώμονε για το κατά πόσο θα πρέπει να μείνει αμετάβλητο το πρώτο τμήμα ή να συμπεριληφθεί διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάγει ανάλογα με την περίπτωση διαφορετικές συνέπειε. Αν ένα κράτο δεν είναι ακόμη μέλο του χώρου Σέγγεν και η έκβαση τη αξιολόγηση είναι αρνητική, ε, η συνέπεια είναι ότι δεν έρεται ο έλεγχο στα σύνορα. Οπότε φτάνουμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση που βρίσκεται στην καρδιά τη συζήτηση και για την οποία συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρακολούθηση, δηλαδή να έχουμε αποτελεσματικά μέσα για να διορθώσουμε κάποιε αδυναμίε, για να εφαρμόσουμε τι συστάσει, αν διαπιστώσουμε κάποιε αδυναμίε, να έχουμε στη διάθεσή μα τα εργαλεία για να τις καλύψουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της έχει προτείνει μια διαδικασία name and shame, δηλαδή να κατανομάζεται ο υπέτειος ώστε με διαφάνεια να ενημερώνονται όλοι και να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για την σωστή εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να διερευνήσουμε και άλλους μηχανισμούς και εργαλεία για τα κράτη-μέλη. Αν θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να θεσπίσουμε και κυρώσεις για το για την καλύτερη παρακολούθηση. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και τη συνέχιση της συζήτησης και είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε και δυνατότητα περαιτέρω κυρώσεων. Σε ό,τι αφορά το τρίτο ζήτημα, την τρίτη ερώτηση, την ε, επέκταση της αξιολόγησης και σε άλλους τομείς, την αξιολόγηση της αμοιβέ εμπιστοσύνη, για παράδειγμα. Δηλαδή, για να διαπιστώσουμε αν κάποιο κράτο μέλο όντω ε, καταπολεμά αποτελεσματικά τη διαφθορά ή αν έχει μέτρα ε, πάταξης του οργανωμένου εγκλήματο. Εδώ επανέρχομαι στο κεκτημένο του Σέγγεν. Τα ιδρυτικά μέλη και μετά τη συμπερίληψη του κεκτημένου Σέγγεν και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το Συμβούλιο προ... ανέπτυξε περαιτέρω το κεκτημένο του Σέγγεν. Τι είναι όμω το κεκτημένο Σέγγεν? Είναι τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα το Συμβούλιο προκειμένου να άρει του ε, ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα ή να κρατήσει ένα χώρο χωρί ε, εσωτερικού ελέγχου. Το Συμβούλιο μιλάει για το αν ένας μηχανισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σέγγεν ή όχι. Αν το Συμβούλιο θεωρήσει ότι ο ένας μηχανισμός εμπίπτει αυτό το κεκτημένο το, για να και θεωρεί ότι μπορούν να έρονται οι έλεγχοι, αυτό το νόημα έχει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αφορά το κεκτημένο του Σέγγεν. Αν θέλουμε να την επεκτείνουμε, θα πρέπει να δούμε τι είδους κεκτημένο θα καλύψει ή το επιπλέον κεκτημένο να χαρακτηριστεί και αυτός κεκτημένο Σέγγεν για να έχει νόημα η επέκταση της αξιολόγηση και σε αυτό. Αυτά ω προ τι τρει ερωτήσει που θέσατε και περιμένω τη συνέχιση των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση τώρα. Έχω έναν κατάλογο των συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Κύριο Σέντσιου πρώτος. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους εμπειρογνώμονες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κάρλος Κοέλιο. Είναι ένα ειδήμων ε, στον ε, κλάδο του και εγώ ως ε, σκιώδης εισηγητής ε, της έκθεσής του υποστηρίζω αυτά τα οποία λέει. Εγώ έλαβα πολλές ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Κοέγιο. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε επίσης αυτό το διπλό σύστημα αξιολόγησης για τις υποψήφιες χώρες. Η πρόταση για την εφαρμογή του, ε, του Frontex είναι πολύ θετική και η πρόταση της Γαλλίας για το νέο σύστημα αξιολόγησης για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, τι μπορώ να πω. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι καλά, αλλά πρέπει όμως να τα ορίσουμε πρώτα και να δούμε τι θα καλύπτουν γιατί πάντα μπορεί να τα χρησιμο... αυτά τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικές σκοπιμότητες. Εμείς πρέπει να σταθεροποιήσουμε το κεκτημένο του Σέγγεν από τεχνικής πλευράς. για να δούμε πόσοι λαθρομετανάστες πέρασαν τα σύνορα ή πόσα, ε, πόσες κλοπές ε, γίνανε, ε, χρειάζονται τεχνικές μέθοδοι. Και όσες χώρες έχουν ξεπεράσει πια αυτό το επίπεδο αξιολόγησης σε νομικό επίπεδο θα πρέπει να γίνουν πλήρη μέλη. Τώρα για τις κυρώσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται προοδευτικά και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την βαρύτητα των διαφόρων παραβιάσεων και θα πρέπει να υπάρχουν και τα συστήματα και συστήματα βοήθειας για αυτούς που δεν σεβάστηκαν τα κριτήρια Σέγγεν διότι δεν η αθέτηση των όρων Σέγγεν πολλές φορές ε, μπορεί να οφείλεται σε ζητήματα που δεν εξαρτώνται από τη θέληση των κρατών μελών. Ένα άλλο σημείο είναι ότι δεν θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να παρακολουθεί ως θεατής τα διαμοιβόμενα στο Σέγγεν. Η Λισαβόνα μας δίνει πλήρες, αρμοδιο... πλήρες αρμοδιότητες και το Κοινοβούλιο θα πρέπει και αυτό να ενημερώνεται και για τους όρους επίσκεψης και για τους όρους αξιολόγησης. Και πρέπει και εμείς να εμπλακούμε σε αυτήν τη διαδικασία για να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είχαμε πρότινος όταν μιλούσαμε για την αξιολόγηση των εκθέσεων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στο Σέγγεν. Ο κύριος Σίλτσεφ. Благодаря, господин председател. Аз също искам Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κοέγιο, και εγώ με τη σειρά μου και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Σήμερα συζητούμε ε, τη πολύ ωραία πρόταση του κυρίου Κοέγιο ε, αλλά ακούσαμε και εμπειρογνώμονες από τη Γαλλία και την Τσεχία που προσπαθούν και εκείνοι να δώσουν μια νέα πνοή σε αυτό το νέο οικοδόμημα. Ελπίζω σήμερα να αποκτήσουμε μια θεώρηση και ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο θα λύνουμε τα προβλήματά μας στο μέλλον. Ε, και ο εισηγητής κάνει προσπάθειες και οι για να ξεπεράσουμε κάποιες ε, προκαταλήψεις ε, σχετικά με την εισδοχή της ε, Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην επικείμενη στο Σέγγεν και θέλουν να προσθέσουν και εγγυήσει ότι αν μπουν αυτές οι δύο χώρες στο Σέγγεν δεν θα σημαίνει μεγαλύτερη απειλή ή περισσότερα προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβάθμιση λέτε του μηχανισμού αξιολόγησης. Και εγώ θέλω βελτίωση αυτού του μηχανισμού. Έτσι το είπε και ο κύριος Κοέγιο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ένας προηγμένος μηχανισμός. Να μην πιστεύει ο κόσμος ότι θα επιπλέξουμε το μηχανισμό, αλλά θα το βελτιώσουμε έτσι ώστε η... δηλαδή δεν θα είναι ένας ε, μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Όχι. Αυτό που θέλουμε να βελτιωθεί, να τελειοποιηθεί ε, και όχι να ε, γίνει πιο αυστηρός ή πιο ε, βίαιος αυτός ο μηχανισμός. Κάποιος από τους εμπειρογνώμονες μίλησε για σημαντικές κυρώσεις και ο εκπρόσωπος ε, της γαλλικής πολιτικής σχολής προφανώς ανέφερε ένα σύστημα κυρώσεων. Μεγάλος αριθμός πολιτών και πολιτικών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα προτιμούσαν ένα σύστημα κυρώσεων παρά κάποιες δυνατές κυρώσεις. Γιατί τι θα πει δυνατές κυρώσεις, ενδεχομένως κάποια στιγμή να σου επιβληθούν, αλλά δεν ξέρεις ούτε πότε ούτε κυρώσεις θα αυτές. Αν υπάρχει ένα σύστημα όμως εκ των προτέρων ορισμένο, είναι σαφή τα πράγματα και πολύ πιο δίκαια. Ναι, να μην είναι δυνητικές οι κυρώσει, αλλά πολύ γνωστές εκ των προτέρων και σαφώς καθορισμένες. Και όχι απλώς αυτόματα με κάποιους υπολογιστές, αλλά με κάποια επιπλέον ανάλυση. Γιατί και εμείς από τη συμμετοχή μας και από τον καλό έλεγχο θα έχουμε ωφέλη να αποκομίσουμε. Και σύντομα τα σύνορά μας θα γίνουν και εξωτερικά σύνορα τη Ένωση ω προ το Σέγγεν. Και ερχόμαστε τώρα στο πιο λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει τα διαφορετικά κριτήρια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς εδώ και συγκεκριμένοι. Διότι μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί μια ιδέα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, ίσως να αναφερθούν στη συνέχεια και άλλοι συνάδελφοι σε αυτό. Τι εννοώ. ένα τμήμα του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος θα ε, συμπεριληφθεί στο νέο μηχανισμό αξιολόγησης του Σέγγεν. Ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ως ε, εγχείρημα, ως πείραμα είναι κάπως αμφίβολο, γιατί αν αρχίζουμε να κατηγοριοποιούμε τις χώρες, να τις κατατάσσουμε με βάση τη διαφθορά, με βάση την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, πάντα θα έχουμε διαφωνίες και θα σπέρνουμε αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν κανένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχει κάνει τέτοια ταξινόμηση των κρατών μελών, επίπεδο διαφθοράς ή αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Αυτά το φαινόμενο είναι δυναμικά, εξελίσσονται. Μπορεί να υπάρχει διαφθορά κάλλιστα σε παλιά κράτη-μέλη και σε παλιές δημοκρατίες και να είναι τελείως απούσα ε, στα νέα κράτη-μέλη και το αντίστροφο φυσικά. Ε, λοιπόν, η συνεργασία και ο έλεγχος και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της δικαιοσύνης μπορούν να γίνουν αλλά δεν είναι του παρόντος. Ίσως θα χρειαστεί κάποιος χρόνος γι' αυτό. Διότι οι κοινωνίες μας είναι πρόθυμες με να δουν αυτούς τους μηχανισμούς να ε, ευδοκιμούν και δεν θα πρέπει αυτομάτως να ε, αφαιρούμε κάποια στοιχεία από τον παλιό μηχανισμό και να εντάσσουμε στο καινούριο. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα πετύχουμε στην προσπάθεια αυτή και σήμερα σε αυτό που συζητούμε. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έγιναν πολύ σοβαρές προπαρασκευαστικές ενέργειες και προσπάθειες περασμένους μήνες, επισκέψεις στα βουλγαρο-τουρκικά σύνορα, στις ακτές της Βουλγαρίας και αναφέρθηκε σοβαρή πρόοδος. φαίνεται ότι συζητούμε για θέματα ε, τύπου κάποιων μικρών στρατών που έχουν προετοιμαστεί, είναι ετοιμοπόλεμοι, αλλά δεν, έχουν, δεν έχει χρειαστεί να πολεμήσουν ποτέ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συνταχθούμε στο Σέγγεν, πάντα θα μπορούμε να βελτιώσουμε και με τρόπο σοβαρό και συστηματικό τη δράση μας. Και ε, έχοντας υπόψη τις κυρώσεις. Αλλά να μην μιλάμε για ενδεχόμενες δυνητικές πιθανές κυρώσεις. Όχι, να ένα σύστημα κυρώσεων το οποίο να επιβάλλεται γενικώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρινέσκου τώρα. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους εμπειρογνώμονες για την παρουσία τους. Αλλά έχω μη, ένα μόνο ερώτημα και μερικές παρατηρήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν μόνο σε αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα ή όχι. Διότι αυτό το οποίο αναφέρθηκαν είναι κάτι για το οποίο δεν συζητάμε σήμερα. Εμείς σήμερα μιλάμε για έναν κανονισμό, για τη θέσπιση δηλαδή ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν για το αν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται. Και μόνο για αυτόν τον νέο κανονισμό πρέπει να μιλήσουμε. Και ορισμένα πράγματα που αναφέρθηκαν από τους εμπειρογνώμονές μας και πιο συγκεκριμένα από το Γάλλο προσκεκλημένο είναι άσχετα με το σημερινό μας θέμα. Είναι σαφέστατο στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για έναν κανονισμό για τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης του κεκτημένου Σέγγεν. Και μιλάμε εδώ για θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για το αν εφαρμόζεται το κεκτημένο του Σέγγεν σε χώρες οι οποίες ήδη είναι μέλη του Σέγγεν. Εγώ είμαι σύμφωνος ότι χρειάζονται όμοια κριτήρια για όλες τις χώρες και για τις χώρες που είναι μέλη αλλά και για τις υποψήφιες χώρες. Τα ίδια κριτήρια και για τους δύο. Όμως, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται διαφορετικά. Διότι, πώς θέλετε εσείς να εφαρμόσετε αυτόν τον κανονισμό σε μια χώρα η οποία ήδη πρέπει να εφαρμόζει το κεκτημένο του Σέγγεν. Εδώ μιλάμε για ένα ετήσιο πρόγραμμα, για την ανάλυση κινδύνων. Δεν μπορείτε όμως να εφαρμόσετε τα ίδια κριτήρια σε μια χώρα η οποία είναι απλώς υποψήφια για το Σέγγεν. Διότι αυτή η χώρα χρειάστηκε να περάσει μια μεταβατική φάση που κράτησε 2, 3, 4 χρόνια. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαφορετική. Διότι η χώρα η οποία είναι υποψήφια ξεκινάει από το μηδέν. Αυτός ο κανονισμός αφορά στις χώρες οι οποίες ήδη είναι μέλη του Σέγγεν. Και εκεί εξετάζουμε αν το κεκτημένο του Σέγγεν εφαρμόζεται σωστά. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις, πάλι οι προδιαγραφές δεν θα πρέπει να είναι ίδιες. Οι χώρες οι οποίες δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη του Σέγγεν δεν μπορεί να τιμωρούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τις χώρες που ήδη είναι μέλη του Σέγγεν. Από την απονομική πλευράς κάτι τέτοιο δεν στέκει. Πιστεύω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι σαφέστατα. Τα κριτήρια πρέπει να είναι τα ίδια για όλους, αλλά οι εφαρμοστικές λεπτομέρειες πρέπει να είναι διαφορετικές. Δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε στο ίδιο επίπεδο χώρες που είναι πλήρη μέλη με χώρες υποψήφιες. Πιστεύω ότι οι κυρώσει είναι καλό πράγμα. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα κυρώσεων. Αλλά αυτές οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του κανονισμού, αλλά να ανήκουν στο κεκτημένο του Σέγγεν. Δηλαδή κυρώσεις για όλους όσους δεν σέβονται τα κριτήρια. Εμείς εδώ μιλάμε για μια διαδικασία, για έναν μηχανισμό, ετήσιο ή πολυετή, στη βάση της ανάλυσης των κινδύνων και ορίζουμε αν γίνεται σεβαστό ή όχι το κεκτημένο. Σεβασμός του κεκτημένου και βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία. Και στη συνέχεια Αυτά στέλνονται σε μια επιτροπή βάσει του άρθρου 15. όπου πια το Συμβούλιο αποφασίζει αν θα πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις λοιπόν θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της συμφωνίας της ίδιας Για νέα κριτήρια τώρα. Μπορούμε κάλλιστα να το συζητήσουμε. Αλλά τα νέα κριτήρια και αυτά θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Δηλαδή να το να προσθέτουμε νέα κριτήρια ή να βγάζουμε κριτήρια από την συμφωνία, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί αλλού. Δεν μπορούμε εμείς να συζητάμε εδώ για νέα κριτήρια, διότι είναι εκτός αντικειμένου του κανονισμού του ίδιου. Σίγουρα, εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Κομισιόν, αλλά και των δύο οργανισμών της Frontex και της Europol. Ευχαριστώ. Η ε, Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Είναι ευαίσθητο το θέμα, όντω και λεπτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι αποσκοπούμε. Από τη μια θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, σαφέστατο είναι αυτό. Από την άλλη και διαφύλαξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Αυτά πώς αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν πάντα θα πρέπει να το σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για αξιολόγηση του Σέγγεν και συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αλίμονο, αλλά το θέμα είναι πώς θα διατηρούμε αυτή την ισορροπία. Και για μένα είναι και ένα θέμα διαφύλαξης και κάποιου μέτρου έτσι, και κάποια αναλογικότητας. Γιατί για τις χώρες που θα μπουν ή που μπήκαν ήδη στο Σέγγεν θα πρέπει να υπάρχουν ίδιες υποχρεώσεις και ίδια δικαιώματα και όντω να υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο. Να υπάρχουν κριτήρια εισαγωγή και δυνατότητα διευκόλυνση για τι υποψήφιε χώρε για την ένταξή τους. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να οδηγήσουν παρόλα αυτά σε ένα ενιαίο ε, σύστημα και κατάλογο κριτηρίων και να τηρούμε κιόλα. αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διχαστεί και το λέω πραγματικά έτσι σκληρά συνειδητά. Δεύτερον, η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά το ίδιο το Σέγγεν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το Σέγγεν. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε τι θέλουμε να αξιολογούμε, τι θέλουμε να μετράμε. Και έχω μια ερώτηση ε, στο Γάλλο συνάδελφο. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό πώς μεταφράζεται, τι σημαίνει. Ότι κάθε χρόνο αποκαλύπτονται ε, τόσοι ε, διεφθαρμένοι δήμαρχοι, α πούμε, και αυτό τι θα πει, πώς το μετράμε και τι σημαίνει. Δηλαδή τι ζητάμε. Μήπω είναι και αντιπαραγωγικό καμιά φορά για τη συνοχή ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ελλείμματα τώρα και κυρώσεις. Είχα, ακούσαμε, να σας πω τι ακούσαμε. Ε, αποκλεισμός από το Σέγγεν, αποτρεπτικός μηχανισμός, αναστολή ατασταλίες, παρατυπίες. Ε, προσοχή με τους χαρακτηρισμούς και με τα μέσα. Οι κυρώσεις μπορεί όντω να είναι αντιπαραγωγικές και να πηγαίνουν σε τελείως στρεβλή κατεύθυνση. Προσοχή λοιπόν. Βήμα-βήμα να το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα έχουμε άλλωστε και ευκαιρία γι' αυτό. Αλλά μην λέμε τόσο ελαφρά την καρδία ότι μπράβο αυτός είναι ο σωστός δρόμος και να παταχθούν. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη αυτή η λύση. Και να μιλήσω λίγο για τη Frontex και την Europol. Για, από τη Γερμανία η Frontex ε, είναι εντάξει. Έχουμε θαυμάσια γεωγραφική θέση και δεν έχουμε ε, να ανησυχούμε για ε, τους μετανάστες και όταν έχουμε τη λαθρομετανάστευση έχουμε και καλό μητρό. Ναι, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και την κατάσταση των χωρών που έχουν ιδιαιτερότητες που είναι διαφορετικές από εμά και να υπάρχει ένα περιθώριο ε, χειρισμών και λιγμών. Αυτά προς το παρόν. Έχω να πω κι άλλα, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. κυρία Στάρουκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατη. Μία ερώτηση έχω προς συμπειρογνώμονες για τις κυρώσεις. Είπατε ότι δεν αρκούν οι κυρώσεις γιατί ε, είναι πολύ ασθενής κύρωση επανειλημμένες επισκέψεις. Βέβαια αναφέρατε και την άλλη ακραία κύρωση που είναι ο αποκλεισμό από το Σέγγεν. Εσείς όμως ε, για ποιες κυρώσεις υποστηρίζετε, τι κυρώσεις προτείνετε. Γιατί μας μιλήσατε για τα δύο άκρα αλλά δεν μας είπατε εσείς τι προτιμάτε. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Και μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Τσεχίας. Εκπροσωπείται ένα κράτος ε, που προσχώρησε στο Σέγγεν στην τελευταία διεύρυνση του χώρου Σέγγεν και έχετε διαφορετική εμπειρία φυσικά από τον Γάλλο εκπρόσωπο γιατί εσείς έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από το δεύτερο κύμα της διεύρυνσης ε, Σέγγεν. Ευχαριστούμε κύριε Σδάνοκα. Θα πρότεινα να ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες για μια σύντομη αντίδραση πριν ε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τη δευτερολογία του κύριου Κοέλη. Παρακαλώ, είστε σύντομοι γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Σούστρο, είστε πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι είχα πει αρκετά στην εισαγωγική μου ομιλία και αυτά που είπα προηγουμένως νομίζω ότι καλύπτουν και τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Οπότε θα περιοριστώ σε κάποιους ε, σύντομους σχολιασμούς. Να απαντήσω καταρχήν στον κύριο Ήλτσεφ. Μάλλον με παρεξηγήσατε κύριε Ήλτσεφ. Λυπούμε που δεν ήμουν αρκετά σαφής προηγουμένως. Είπα πιθανές κυρώσεις. Είναι υποθετική αυτή η συζήτηση που έχουμε. Γι' αυτό μίλησα για πιθανές ή δυνητικές κυρώσεις. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Ήλτσεφ ότι αν θέλουμε αποτελεσματική αντίδραση θα πρέπει να θεσπίσουμε και κυρώσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν ξέρω αν θα είναι προληπτικό ή κατασταλτικό το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είναι προβλέψιμο και σαφές. Σε καμία περίπτωση αβέβαιο και δυνητικό. Και θέλουμε στην αξιολόγηση, στο σύστημα αξιολόγησης του Σέγγεν θέλουμε να κρατήσουμε και τα συμπεράσματα του Στρασβούργου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σχόλια του κυρίου Ήλτσεφ, και εμείς διαπιστώσαμε με ικανοποίηση την πρόοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές των δύο χωρών για προσχώρηση στο Σέγγεν. Ως προς τον κύριο Μαρινέσκου, θα ήθελα να πω ότι όντως η... θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι διαφορές μεταξύ του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας και του καθεστώτος της χώρας μέλους του Σέγγεν. Το θέμα των κυρώσεων φυσικά είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο και μόλις τώρα ξεκίνησε η σχετική συζήτηση. και το θεωρούμε ως πραγματικά ίστατη λύση το θέμα των κυρώσεων. Μπορώ να φανταστώ θεωρητικά μια κατάσταση με κύρωση αποκλεισμού ενός ε, κράτους μέλους, αλλά πραγματικά αυτή είναι η ίστατη λύση, η έσχατη λύση. Θα μπορούσα να επαναλάβω μερικές από τις ιδέες που αναφέρθηκαν πριν φτάσουμε σε αυτή την έσχατη λύση, νομίζω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις προηγούμενες ε, δυνατότητες για να διορθώσουμε τα προβλήματα και να καλύψουμε τις αδυναμίες χωρίς να προσφύγουμε σε αυτή την έσχατη λύση που είναι αποφακτέα, που είναι και η πιο βάναυση ε, κύρωση, ο αποκλεισμό δηλαδή. Πάντως και στις μελλοντικές συζητήσεις πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ποιότητα ή την, το βαθμό αυστηρότητας ε, των προτινόμενων μέτρων και να αναλύσουμε την ιδέα για τον ίδιο το χαρακτήρα των δυνητικών κυρώσεων. Όλα αυτά θα αποσαφινιστούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεμπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. όσον αφορά στους, προσανε... στους προσανατολισμούς που υπέδειξα. Μα πρόκειται για κάτι τεχνικό και για την βελτίωση του μηχανισμού χρειάζονται τεχνικές λύσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σέγγεν και όλα γυρνάνε γύρω από αυτό το στόχο. Εμείς ψάχνουμε λύσεις που δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεθούν. Αναφέραμε τη δυσκολία του ορισμού κριτηρίων αξιολόγησης, νέων κριτηρίων εμπιστοσύνης, που να επιτρέπουν στα κράτη Σέγγεν να συνεργάζονται εύρυθμα μεταξύ τους. Και πρόκειται εδώ για μια πρόκληση γύρω από την οποία προβληματιζόμαστε για το πώς εμείς θα αξιολογήσουμε ε, τις ε, υπηρεσίες ε, των <coughs> και μέσα στις στις εθνικές μας υπηρεσίες για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε όλα αυτά και σε επίπεδο δεοντολογίας και με προδιαγραφές ηθικής αυτών των υπηρεσιών που πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Σέγγεν. Αλλά ε, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Και αν δεν, αν δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα επανερχόμαστε συνεχώς στο μέλλον γύρω από αυτά τα θέματα. Και τα θέματα αυτά θα επανέρχονται αν δεν ληφθεί υπόψη και το νομικό πλαίσιο για να βρούμε τις λύσεις. Τώρα εμείς ως εμπειρογνώμονες φυσικά ψάχνουμε τις λύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Ωραία, να ακούσουμε τώρα. Τα συμπερασματικά από τον κύριο Κοέγιο. Πού θα πείτε τελευταία σχόλια πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να κάνω δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Παρατήρηση πρώτη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην συγχαίεται την προσχώρηση της Ρουμανίας και Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν με το νέο σύστημα αξιολόγησης Σέγγεν. Το σύστημα αξιολόγησης Σέγγεν είναι μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απέρριψε τον Οκτώβριο του 2009 μετά από δική μου σύσταση. Ζητήσαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα νέο, ένα νέο σύστημα αξιολόγηση Σέγγεν. Αυτό και έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα αυτό που συζητάμε είναι το μελλοντικό σύστημα αξιολόγηση του Σέγγεν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το νέο σύστημα αξιολόγηση Σέγγεν με την προσχώρηση Ρουμανία και Βουλγαρίας στο Σέγγεν. Μην τα συγχαίρετε λοιπόν, σας θερμοπαρακαλώ. Το γεγονό ότι εξετάζουμε τώρα ένα νέο σύστημα αξιολόγηση Σέγγεν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ω άλοθη η δικαιολογία για να καθυστερήσει η προσχώρηση τη Ρουμανία και Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν. Ούτε μπορούμε να εξετάσουμε το νέο σύστημα αξιολόγηση του Σέγγεν με το φόβο ότι θα εφαρμοστεί σε ορισμένες μόνο χώρες. Γιατί αν τα μπερδέψουμε αυτά τα δύο θέματα θα αλλοιώσουμε τελείως το περιεχόμενο της συζήτησης και θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Παρακαλώ να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της και προσβλέπω σε στενή συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία στη διαδικασία της συναπόφασης. Γιατί αυτή ισχύει για την περίπτωση του νέου συστήματος αξιολόγης έγκαιρ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσω των δύο από της Τσεχίας και της ε, Γαλλίας και τις δύο χώρες, γιατί ούτε η Τσεχική Δημοκρατία ούτε η Γαλλία ανήκαν στη μικρή ομάδα των χωρών που ε, ζήτησαν να παραγωνίσουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομική βάση της εναπόφασης ε, προσπάθησαν να καταρρύψουν αυτή τη νομική βάση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστεί η συναπόφαση. Αλλά ούτε η Γαλλία ούτε η Τσεχική Δημοκρατία ήταν, ε, ήταν τμήματα, ε, ανήκαν σε αυτή την ολιγομελή ομάδα των ε, χωρών μελών που προσπάθησαν να καταρρύψουν το εύλογο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ισχύσει συναπόφαση στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Γαλλία και την Τσεχία που δεν υποστήριξαν τις α, λίγες αυτές χώρες που το ζήτησαν. Νομίζω ότι από τη συζήτηση φάνηκε ότι οι περισσότεροι τάσσονται κατά των διπλών προδιαγραφών και των δύο μέτρων και σταθμών. Θα πρέπει τα κριτήρια να ισχύουν για όλες τις χώρες, είτε είναι αυτές οι υποψήφιες για το χώρο Σέγγεν, είτε είναι ήδη μέλη του χώρου Σέγγεν. Δεύτερον, νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι αν δεν θέλουμε διπλά μέτρα και σταθμά, θα πρέπει να δεχτούμε και τις συνέπειες της αξιολόγησης. Αλλιώς θα, θα εφαρμόζουμε στις υποψήφιες χώρες αρνητική απόρριψη του να εισέλθουν εφόσον είναι αρνητική αξιολόγηση, αλλά για τις χώρες που είναι ήδη μέλη η αρνητική αξιολόγηση δεν θα έχει καμία συνέπεια. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Οι περισσότεροι συναδέλφοι είπαν ότι πριν την επιβολή κυρώσεων καλό θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε τις χώρες να λύσουν τα προβλήματά τους και όχι αμέσως να προσφύγουμε στις κυρώσεις. Συμφωνώ. Στην τελική φάση όμως, αν μια χώρα δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσει ε, των κανόνων ασφαλείας στο χώρο Σέγγεν και είναι ήδη μέλος του χώρου Σέγγεν, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Πάντως συμφωνώ ότι πρώτα θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήματα και σίγουρα να ισχύουν οι ίδιες κυρώσεις για όλους και όχι δύο μέτρα και σταθμά να μην έχουμε χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Τρίτον, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά και τα νέα κριτήρια. Γιατί υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ανάγκης θέσπισης νέων κριτήριων. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε λεπτομεριακά όλα αυτά τα νέα κριτήρια. Γιατί αν θεσπίσουμε νέα κριτήρια, θα πρέπει αυτά να είναι αντικειμενικά. Για να μην ε, υπάρχει περιθώριο υποκειμενικότητα μεροληψίας που θα αλλοιώσει το σύστημα αξιολόγησης έγκαιν. Και φυσικά, αν θεσπίσουμε νέα κριτήρια, αυτά θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη και τα υποψήφια και τα μέλη και όχι μόνο σε ορισμένα κράτη. Θα ήθελα επίσης να υπογραβεί μισό αυτό που είπε ο κύριος Έντζιου, την ανάγκη να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση του νέου συστήματος αξιολόγησης και να λαμβάνει σωστή ενημέρωση για τις αξιολογήσεις που γίνονται στα σύνορα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα και θέλει να γνωρίζει τι συμβαίνει για να μπορεί να ενημερώσει τους πολίτες και να, πει, να τους πει και να τους πείσει ότι ο χώρος του Σέγγεν είναι ένα ασφαλής χώρος για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, κάτι που επιθυμούν άλλωστε και οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέγιο. Το σχέδιο έκθεσης προβλέπεται να κατατεθεί ε, στη συνεδρίασή μας στις 11 και 12 Απριλίου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους δύο ε, εμπειρογνώμονες, τους αποχαιρετούμε. Και περνάμε μέσω στο επόμενο. Γιατί έχουμε και καθυστέρηση λίγο χρονική και πρέπει να επιταχύνουμε αν θέλουμε να προκάνουμε. Να καλύψουμε όλη την ημερήσια διάταξη για σήμερα. So, we move 15. Συνεχίζουμε. Σημείο 15 συνολική προσέγγιση τώρα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλαγή απόψεων. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων σημειωτέων του εγγράφου εργασία. Είναι ιδέα πρωτοβουλία η έκθεση. Εισηγητή ο φίλο συνάδελφο Άξελ Φω. Θα του δώσουμε το λόγο να μα παρουσιάσει το έγγραφο εργασία και στη συνέχεια ε, θα ανοίξει συζήτηση με συμμετοχή των συναδέλφων και αν θέλουν ε, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο Θα ήθελα όντως να ρίξω μια ματιά στην προστασία των δεδομένων, μια νέα ματιά, μια φρέσκια ματιά. Τι χρειάζεται σήμερα δηλαδή. Και θα ήθελα να κάνω και μια διαφήμιση, να ζητήσω έναν επαναπροσανατολισμό. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Οι εξελίξεις των τελευταίων 15-20 ετών δείχνουν ότι η ψηφιακή εποχή έχει αναπτυχθεί παγκοσμίω με τέτοιο τρόπο που η οικονομία, η ασφάλεια, οι επικοινωνίες, συγγνώμη, ο πρόεδρος διακόπτη. Παρακαλούνται όσοι αποχωρούν ε, να αποχωρούν ησύχως για να ακούμε εμείς τον εισηγητή. Λοιπόν, έλεγα ότι ε, όλοι οι τομείς της καθημερινής και της ιδιωτικής μας ζωής επηρεάζονται και ζούμε ε, σε μια εποχή που χωρίς συλλογή δεδομένων, χωρίς ε, αποθήκευσή τους και ύπαρξη δεδομένων καν είναι αδιανόητη. Είναι τέτοια τεχνολογία. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς ε, σου παίρνουν τα δεδομένα, τα στέλνουν δεξιά και αριστερά και ζούμε επίσης και το εξής. Οι νέοι ακριβώς ε, που συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τα προσωπικά του στοιχεία με τρόπο έτσι πολύ επιπόλαιο, φωτογραφίες, βγάζουν ε, αβίαστα. Ε, και αυτό θέτει και ένα ερώτημα, το πώς προστατεύει ο καθένας τα προσωπικά του δεδομένα και την ιδιωτική του ζωή στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν <coughs> δεν μπορεί πια κανείς να ελέγχει τι δεδομένα υπάρχουν για τον καθένα μας, ειδικά στο διαδίκτυο και επίσης δεν μπορούμε να ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά, ποιος τα διαβάζει καν. Ε, γι' αυτό λοιπόν η σημερινή προστασία δεδομένων όλο και περισσότερο ε, έχει να υπομειστεί ένα βαρύ καθήκον. Γιατί η συλλογή των δεδομένων, η ανάλυση τους, μέχρι και το εμπόριο με τα δεδομένα ή και η κατάχρηση και η ε, πλαστογράφηση ε, και δυνατότητα εντοπισμού και profiling ε, έχουν προσλάβει τεράστιες διατάξεις, διαστάσεις. Συγγνώμη. Και ε, αλλάζει και η προοπτική, θα το χαρακτήριζα έτσι. Στο παρελθόν τα θεμελιώδη δικαιώματα έλεγαν ότι θα πρέπει να προστατεύουμε το μεμονωμένο πολίτη από το κράτος, ενώ σήμερα βλέπουμε το αντίθετο. Ότι το Αυτό που πρέπει να προστατεύουμε είναι τον ιδιώτη από άλλους ιδιώτες που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του. Και σήμερα ο κόσμος μας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ψηφιακή επεξεργασία και ε, μετά βίβαση δεδομένων. Αυτό είναι από τον έλεγχο της αέριας κυκλοφορίας, υγεία, οικονομία, υποδομές, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Όλα αυτά σήμερα ε, μπαίνουν σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική και Οπότε μπαίνουμε ε, σε αυτό το μέσο του μέλλοντος, θα αφήνουμε πίσω μας ψηφιακά χνάρια και θα μπορούν να μας εντοπίζουν, να μας ανοιχνεύουμε βάσει τα ίχνη μας. Και τώρα μιλάμε για ευφυή ψυγεία. Για ευφυή δίκτυα ηλεκτρισμού. Θα αφήνουν λοιπόν και ηλεκτρονικά ίχνη και θα, θα φαίνονται οι συνήθειές μας, ε, ε, θα καταγράφονται ηλεκτρονικά και οι καταναλωτικές και τι τρώμε και τι μας αρέσει και πώς ζούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το χειρισμό αυτών των ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών και τη ε, χρήση και κατάχρηση καμιά φορά. Και τονίζω ότι η διευθύνη ευθύνη όλων των συμμετεχόντων σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρώτο απαιτούμενο. Η σημερινή προστασία δεδομένων τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τώρα. Μια σύγχρονη προστασία για μένα και ευφυής θα πρέπει να ε, έχει μια ισορροπία μεταξύ ε, της ατομικής ελευθερίας, της συλλογική ασφάλειας, της αυτοδιάθεσης του καθενός ως προς τις πληροφορίες που διαθέτει σε όποιον θέλει και επίσης και η αναγνώριση ότι μια γρήγορη και αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων είναι εκ των όνων κάνευ σήμερα για να εγγυόμαστε την ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική. Γι' αυτό λοιπόν οι αρχές προστασίας δεδομένων σήμερα θα πρέπει να προσανατολίζονται στα μεμονωμένα ε, συμφέροντα και μελήματα του κάθε ιδιώτη και πολίτη, αλλά και η οικονομία χρειάζεται στοιχεία ε, και δεν μπορεί να εμποδίζεται. Ε, βεβαίως και το διαδίκτυο ολόκληρο δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Ε, θα πρέπει να προσανατολισόμαστε στο τι είναι εφικτό, τι είναι δυνατό, αλλά το κράτος έχει διοικητική ευθύνη να σέβεται και να προστατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και, και τη γενική ασφάλεια. Λοιπόν, για μένα για να έχουν επιτυχία αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να δούμε αν καταφέρουμε εμείς στο μέλλον να έχουμε μια προστασία των Ευρωπαίων πολιτών ανεξάρτητα από το που εδρεύει κάθε εταιρεία ή ε, ο σερβερ ε, να μπορεί καθένας να προσφεύγει και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Και επίσης θα ήθελα να πω τι σημαίνει η προστασία των δεδομένων σήμερα για τους πολίτες και για τη βιομηχανία, για την οικονομία. Είναι πολύ σημαντική η προστασία των δεδομένων σήμερα και για την προστασία των πολιτών και για την προστασία της οικονομίας. Είναι ευρύτατη η χρήση του διαδικτύου και επειδή είναι και θα παραμείνει το μέσον του μέλλοντος, προσλαμβάνω όλο ιδιαίτερη σημασία και τα μέσα αυτά, όλα αυτά στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Λοιπόν, συμπέρασμα. Τι ζητώ να έχουμε ένα νέο δίκαιο προστασίας δεδομένων ε, για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας το παρουσιάσω αυτό με τρία διαφορετικά σημεία. Το επίπεδο ασφαλείας που θέλουμε και προστασίας καλύτερα να εγγυηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι το ίδιο, στρεβλώνει αυτό τον ανταγωνισμό στην εσωτερική ε, ε, αγορά και ξυλώνει, ξεφτίζει η προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν έχουμε υπόψη μας ένα νομικό μέσο που θα εξασφάλιζε υψηλές προδιαγραφές και ενιαίες, αυτό είναι κανονισμός. Ενδεχομένως θα το δούμε αυτό με τους εισηγητές. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος, να είναι ενιαία η προστασία παντού το ίδιο. Οι ίδιες προδιαγραφές, το ίδιο επίπεδο, αλλιώς δεν γίνεται εσωτερική αγορά. και πέρα από την Ένωση και τελικά να έχουμε μια πλήρη εναρμόνιση που να πούμε κανένα κράτος δεν επιτρέπεται να θεσπίζει προδιαγραφές υψηλότερες ή χαμηλότερες. Το ίδιο θα ίσχυε για μένα αν συνδέαμε την προστασία των δεδομένων με κάποια πρόσωπα. Δηλαδή κάπου στον κόσμο υπάρχει μια εταιρεία που χειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα. Αυτό θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ως προς το εξής. Όποιος χρησιμοποιεί δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών εντάσσεται ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή ακόμα και εταιρείε που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά επεξεργάζονται ε, στοιχεία και δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών υπόκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Να δούμε πώς αυτό θα γίνει στη συνέχεια δυνατό να προσβάλλεται σε δικαστήρια. Έτσι, γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλα. Και ο καθένας από εμά θα κληθεί στο μέλλον να αντιδράσει ανάλογα και στα κράτη-μέλη να το επιβάλλουμε και να τηρείται με τρόπο ενιαίο. Προσέχοντας πάντα ε, ότι θα εφαρμόζεται. Κάτι άλλο βέβαια θα το συζητήσουμε και αργότερα, δεν θα λήξει εδώ. Ε, αυτό καθιστά περιττή τη συμφωνία του Safe Harbor, του ε, ασφαλούς λιμένος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τέτοια συμφωνία, ιδιαίτερα τη στιγμή που θεωρούμε ότι δεν ε, λειτουργεί σωστά, μήπως να την καταργήσουμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή και περίπλοκη, αλλά και στον ανταγωνισμό έχουμε τα ίδια με τις αρχές ε, ανταγωνισμού και καταπολέμηση των καρτέλ και των ολιγοπολίων. Ένα τρίτο για την ενιαία εφαρμογή ενός δικαίου για την προστασία των δεδομένων. Προσπαθήσουμε να εντάξουμε εδώ τον παλιό τρίτο πυλώνα, αν θυμάστε. Και να φτιάξουμε μια ρύθμιση που να ισχύει ευρέως. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις ιδιαίτερότητε και σε όλες τις λεπτομέρειες, έτσι κι αλλιώς ένα κανονισμό δεν γίνεται, αλλά τουλάχιστον να θέσουμε τα θεμέλια, τις αρχέ στον κανονισμό και από εκεί και πέρα για τον τρίτο πυλώνα μπορεί να χρειαστεί κάποια έκτακτη μορφή, ένα ειδικό νομικό μέσο, δεν ξέρω. Επίσης, πού θα πρέπει να προσανατολιστούμε αν έχουμε ένα επίπεδο αξιών, ας πούμε, ή θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα πρέπει να προσανατολισόμαστε στην ελευθερία, στην αυτοδιάθεση, αλλά και στην ίδια ευθύνη του καθενός από εμάς. Και στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει μια αρχή, η επιταγή της... Ε, ε, να καταλαβαίνει κανείς, να έχει συνέστηση, να έχει επίγνωση ε, το τι ε, συνέπειες θα έχουν οι πράξεις του. Και αυτό δηλαδή δίνει ιδιαίτερη ευθύνη σε όλους εκείνους που ασχολούνται με δεδομένα προσωπικά. Αυτό αρχίζει από το ίδιο το άτομο. Όταν κάποιος κάνει κάτι φέρει και την ευθύνη γι' αυτό. Και θα πρέπει να την έχει ε, συνειδητοποιημένη αυτή την ευθύνη. Και αυτό ισχύει για τους providers από εκεί και πέρα και κάποιους άλλους που συλλέγουν στοιχεία και τα χειρίζονται. Ότι είναι Ιδιαίτερες οι ευθύνες περιγράφονται και ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό έχει και ευθύνες για όλους. Έρχομαι τώρα στα συγκεκριμένα. Από πλευράς δικαίου τώρα για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων και δεδομένων. Συγγνώμη. Αν επιλέξουμε αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της συγκατάθεσης, γιατί δεν ξέρουμε ποια στοιχεία μαζεύει ποιος, για ποιο σκοπό και πόσο χρόνο τα αποθηκεύει και πού. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που συλλέγουν δεδομένα και προσωπικά τα δικτυώνουν, τα συνδυάζουν χωρίς να έχουν καν την άδεια να το κάνουν. Δηλαδή και πάλι εδώ πρόκειται για τόνωση των δικαιωμάτων του καθενός και προσωπική ευθύνη θα πρέπει ο ιδιώτης να έχει εκείνος τον έλεγχο το ποιο χρησιμοποιεί και με ποιο τρόπο τα δεδομένα που τον αφορούν. Και να μπορεί και να προσφεύγει κάπου. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στην καθημερινή ζωή, δηλαδή όχι την επικραμμική, offline, να μεταφερθούν όλα αυτά και online να είναι κύριος των δεδομένων του ο κάθε άνθρωπος. Και όταν κάποιος ε, τα χρησιμοποιεί και τα, τα χειρίζεται θα πρέπει ε, να έχει δώσει ο ενδιαφερόμενος τη συγκατάθεσή του ρητά και, και ξεκάθαρα. Κάτι άλλο που συνδέεται πάρα πολύ με αυτό είναι η αρχή της διαφάνειας και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε κατά τη γνώμη μου αύξηση της διαφάνειας γιατί θεωρώ ότι ο χρήστης θα μπορεί να πρέπει να βλέπει ποια προσωπικά του δεδομένα έχουν αποθηκευτεί και να ζητάει και δια νόμου να μπορεί να απαιτεί να ε, σβήνονται αυτά, να μην αποθηκεύονται. Άλλη αρχή, τρίτη, είναι Τι σκοπό έχει αυτή η συλλογή ε, δεδομένων και θα πρέπει να έχουμε μία φιδό στη διαχείριση και στην κυκλοφορία αυτών. Και ένα τελευταίο. Έχω την αίσθηση ότι η προστασία των δεδομένων δεν είναι κάτι που μπορεί να αναπτυχθεί πάντα για όλους τους ενδιαφερομένους με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί άλλε να είναι οι δραστηριότητες των ιδιωτών εκτός διαδικτύου και άλλες δραστηριότητες των εταιριών. Ή δεν μπορεί ε, ο κόσμος, ο, μη ψηφιακός, ο, ο πραγματικός να μεταφέρεται 100% πάντα κατά απόλυτη αναλογία και αντιστοιχεία και στο διαδίκτυο. μπορεί να χρειάζεται κάποια έκτακτη ρύθμιση, ειδική ρύθμιση ε, για ορισμένα στοιχεία, αλλά σε κοινό πάντα πλαίσιο. Σύντομα, ε, θέλω να σας πω ότι θέλω και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, ελάχιστες μεν, αλλά να ισχύουν παντού, σε όλους τους τομείς καθολικά. Δηλαδή, ε, ενεργητική συγκατάθεση, υποχρέωση ενημέρωσης, δικαίωμα ενημέρωσης, ε, δικαίωμα διόρθωσης καμιά φορά, προστασία των δεδομένων στην επεξεργασία, ε, αξιώσεις ε, αποζημίωσης σε περίπτωση καταχρήσεων, διάρκεια αποθήκευσης, πότε επιτρέπεται η διαβίβαση σε τρίτους, υποβολή και μηνύσεων όταν υπάρχει λόγος και ασφάλεια δικαίου. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, μάλλον θα πρέπει να τα πω πιο σύντομα, αλλά έχω ένα ολόκληρο κατάλογο θεμάτων που θα πρέπει γενικά να μας απασχολήσουν και να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στον επιγραμμικό κόσμο σε αντίθεση με τον πραγματικό ε, δικαίωμα ε, πνευματικό ας πούμε στα εικόνες, φωτογραφίες το δικαίωμα που έχει κάποιος να ξεχαστεί ε, right to be forgotten λέγεται αυτό ε, privacy by design ή privacy by default ότι τα προγράμματα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ιδιωτική σφαίρα τι γίνεται με τα παιδιά, τι γίνεται με τους ανηλίκους, τους εφήβους, ποια είναι προσωπικά δεδομένα, η διεύθυνση IP είναι προσωπικό δεδομένο. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που κανονικά δεν θα πρέπει πάντα να επιτρέπονται τα πάντα, κάποιοι άλλοι τομείς που θα πρέπει να επιτρέπονται ε, για να υπάρχει μια προστασία και στον κόσμο των υπολογιστών και τελειώνω σιγά σιγά. Να σας πω τα εξής τέσσερα ακόμα. Εκτός από τους ορισμούς, όχι μόνο ότι είναι προσωπικά δεδομένα και επειδή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και το cloud computing να πω ποια τα συνοδευτικά μέτρα εντάξει είπαμε διάθεση, ελεύθερη επιλογή, συγκατάθεση από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και οι πολίτες να είναι σε θέση να τα ξέρουν όλα αυτά, να τα γνωρίζουν και να είναι ενήμεροι. Για μένα πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση ως συνοδευτικό μέτρο. Να γνωρίζει ο πολίτης ε, όλα αυτά που τον αφορούν και η θελούσια πιστοποίηση, αν θέλετε, η αυτορύθμιση των εταιριών σε όλους αυτούς τους τομείς όπου ουσιαστικά από πλευράς δικαίου ή πολιτικής δεν μπορούμε κάθε φορά να εκτιμούμε την κατάσταση. Εκεί θα πρέπει να δείχνουν ευθύνη οι διάφοροι κλάδοι των ε, επιχειρήσεων, των διαδικτυακών και επίσης να δούμε πώς θα ελέγχουμε όλα αυτά τα πράγματα. με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων να έχουν σαφή κατάλογο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Και στη μεταφορά στην πράξη να γίνει αυτό που κάνουμε στις αρχές ανταγωνισμού για τα καρτέλ. Σταματώ εδώ προς το παρόν, ελπίζω να σας έδωσα μια καλή εικόνα έτσι, μια επισκόπηση όλων αυτών των ε, πραγμάτων που λέει και το έγγραφο εργασίας και έχω την αίσθηση ότι έχουν νόημα για μια σύγχρονη ε, και λογική προστασία το δεδομένο. και με χαρά περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο προσκεκλημένους, τον Γενικό Διευθυντή Μανσαρβίση και την Γενική Διευθύντρια Λεμπάγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα μας ενημερώσουν για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Αυτό το θέμα αφορά την ανακοίνωση Επιτροπής. Γι' αυτό προτείνω να ακούσουμε και τους συναδέλφους που θέλουν το λόγο, αλλά μια και σε 10 λεπτά θα έρθουν ε, οι δύο γενικοί διευθυντές. Καλό θα ήταν να τους δώσουμε και το λόγο. Πρώτα η κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική γιατί ο εισηγητής μας κάλυψε τα περισσότερα σημεία και τον ευχαριστώ θερμά για το έγγραφο εργασία του. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, δεν είναι φραγμός, δεν είναι εμπόδιο στη ροή των δεδομένων. Αντίθετα, είναι προϋπόθεση για ελεύθερη ροή δεδομένων. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το ζητούμενο για μας. Συμφωνώ με τον εισηγητή και έχω την αίσθηση ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα εκεί οδεύει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα νέο μηχανισμό ή ένα νέο πλαίσιο για την προστασία δεδομένων που θα καλύπτει όλες τις χρήσεις προσωπικών δεδομένων, είτε για εμπορικούς σκοπούς, είτε για ε, λόγους δικαιοσύνης, εφαρμογής δικαιοσύνης και θα γίνεται μια ενοποίηση των μηχανισμών που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πρώτο και τρίτο πυλώνα. Η εναρμόνιση είναι ένα άλλο νευραλγικό σημείο και για τους πολίτες αλλά και για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ε, σοβαρές δυσκολίες γιατί οι προδιαγραφές και οι κανόνες είναι διαφορετικές στις χώρες μέλη, οπότε προβληματίζονται πώς ε, να τις στηρίσουν οι επιχειρήσεις. Καλό θα ήταν να έχουμε ένα ενιαίο, διαφανές και εναρμονισμένο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διευκολύνει πολύ και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Άρα, μάλλον ε, κανονισμός θα ήταν το πιο κατάλληλο εργαλείο παρά οδηγία. Θα δούμε τελικά. Πάντως, ό,τι κατεύθυνση και αν ακολουθήσουμε και ό,τι νομοθετικό μέτρο και αν υιοθετήσουμε, θα πρέπει το μέσο αυτό να είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη και θα μας εξυπηρετήσει στο μέλλον, γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ότι ο ρυθμός νομοπαρασκευής. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ενισχυθούν και οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χθε είχα κάνει μια πρόταση στα πλαίσια της συζήτησης του SWIFT, αλλά καλό θα ήταν να εξετάσουμε γενικότερα, να επιβάλλουμε δηλαδή αυστηρές κυρώσεις σε εκείνους που καταχρώνται των προσωπικών δεδομένων, ακόμη και ποινικέ ε, κυρώσεις, δηλαδή να σε ακραίε περιπτώσει, σοβαρή παραβίαση να επιβάλλονται ακόμη και ποινέ. Νομίζω ότι δύο είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι πολύ δύσκολες. Η πρώτη πρόκληση είναι να νομοθετήσουμε για συγκεκριμένη επικράτεια όταν τα δεδομένα δεν προορίζονται για αυτή την επικράτεια και χαίρομαι που χθε η Επίτροπος Ρέντινγκ ανέφερε ότι δεν θα είναι καθόλου άτολμη και ε, επιφυλακτική, αλλά θα είναι πολύ φιλόδοξη και μαχητική σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Και τέλος έχουμε πολύ σημαντική πρόκληση, γιατί πολύ συχνά μιλούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχουμε συνήθως κατά νου ένα είδος δεδομένων. Η μία δέσμη δεδομένων. Έχουμε κανόνες για την ασφάλεια, για τους ε, στόχους, για τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Πολύ συχνά όμως δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα που θα πρέπει να τύχουν προστασίας, αλλά είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να εμφανιστεί αυτή η προστασία. Και σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Γιατί μερικά δεδομένα μπορεί να είναι ανώδυνα σε, σε, α πλαίσιο και να είναι πολύ επικίνδυνα σε β' πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που πολύ εύκολα θα τις εκμυστηρευτώ σε ένα φίλο, αλλά δεν θα ήθελα να τις μάθει ο εργοδότης μου για παράδειγμα. Οπότε οι βάσει δεδομένων συνήθως δεν απαρτίζονται από ένα είδος δεδομένων. Το θέμα είναι ότι τα συνδυάζονται. Α, ο, καινούργια πρόεδρος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και θα ολοκληρώσω. Αν δηλαδή επιτρέψουμε τη χρήση ενός ε, ε, είδους δεδομένων για ένα σκοπό και ε, επιτρέψουμε άλλο είδος δεδομένων χρήση τους για άλλο σκοπό, Μπορεί να έχουν πέντε τις διαφορετικές αποφάσεις, αν όμως συνδυαστούν αυτά τα δεδομένα για profiling ή για εμπορικούς σκοπούς ή για τις υπηρεσίες, ουσιαστικά δεν έχουμε επιτρέψει τη χρήση αυτού του, του συνδυασμ, των συνδυασμένων δεδομένων. Αλλά τι γίνεται αν αυτό το προφάιλ, αυτά τα συνδυασμένα δεδομένα χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία, για παράδειγμα. Οπότε δεν μα ενδιαφέρει να έχουμε ειδικού κανόνε για συγκεκριμένα είδη δεδομένων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τι προσωπικέ πληροφορίε, τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο βέβαια. Και αδειμονώ για τη στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδης. Ευχαριστούμε, Σόφη. Έχουμε αρχίσει και μένουμε πίσω στο χρονοδιάγραμμα της απογευματινής συνεδρίασης. Δεν είναι και πολύ θετική στιγμή που ανέλαβα την Προεδρία. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Ο κύριος Λαμπρινίδης και μετά Άλβαρο, Άλμπρεχτ, και τελευταία η κυρία Έρνστ. Ελπίζω να εξαντλήσαμε έτσι τον κατάλογο των αγορητών. Ο κύριος Λαμπρινίδης. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη αρχή που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά είναι μπροστά παντού και πολύ πιο εύκολα, ε, επειδή φτάσαμε στην ηλεκτρονική εποχή, ε, οποιαδήποτε αναθεώρηση της του 94-46 θα πρέπει να ενισχύει τους κανόνες για την ιδιωτική ζωή. Και η προσπελασιμότητα θα πρέπει αυτόματα να σημαίνει ότι ε, μένουμε τα χέρια σταυρωμένα ή μένουμε ανήμποροι. Οπότε η αναθεώρηση 95-46 δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των αρχών της, αλλά αντίθετα ενισχυμένη εφαρμογή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της, αλλά και τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας του. Η δεύτερη αρχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω και που θα πρέπει να έχει εφαρμογή εδώ είναι το γεγονός ότι η προστασία των δεδομένων και η οδηγία που θα αναθεωρήσουμε τώρα θα πρέπει να αποτελεί γενική αρχή και θεμελιώδης δικαίωμα. Και στην αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει να ισχύει ισότιμα για όλους. Φυσικά χρειαζόμαστε βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις και ήδη τι έχουμε θεσπίσει σε άλλε νομοθετικέ πράξει, αλλά θα πρέπει οι εξαιρέσει αυτές να είναι περιορισμένε, ανάλογε με το σκοπό, να μπορούμε να καταπολεμήσουμε οργανωμένα έγκλημα κτλ, να εξυπηρετήσουμε του στόχου μα, αλλά οι εξαιρέσει αυτές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο τη οδηγία, αλλά θα πρέπει όντω να είναι εξαιρέσει και να μην γίνουν κανόνα. Επίση, η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να ισχύει για όλου και να έχει τύχει οριζόντιας εφαρμογής. Το θέμα της συνένεσης αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και από τη Σοφία Ιντφέλτ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της συνένεσης. Δεν μπορούμε τώρα στην έκθεσή μας και στην αναθεωρημένη οδηγία ε, για την προστασία δεδομένων δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε ώρες λεπτομέρειες. Πάντως οι θεμελιώδεις αρχές είναι ότι θα πρέπει να είναι ρητή η συνένεση και όχι τεκμαρτή. Συμφωνώ με αυτό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το σημείο στην έκθεση. Δεν θα πρέπει να υπονοείται η συνένεση, αλλά είναι να είναι πραγματικά ρητή. Τώρα, τι είδου ε, μηχανισμό χρειαζόμαστε. Έχουμε το θέμα της εναρμόνιση, γιατί σήμερα και οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες αρχές, οι κυβερνητικές αρχές πολλές φορές ε, καλούνται να εφαρμόσουν διαφορετικές προδιαγραφές, διαφορετικούς κανόνες και αυτό είναι κακό και για τις επιχειρήσεις και για την προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και για την αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία. Πολλοί θα τάσσονταν μάλλον υπέρ του κανονισμού, αλλά θα έλεγα ότι αν ο κανονισμός ε, όντως μιλάει για, το μέγιστο κοινό παρανομαστή, εντάξει, αλλά αν ευθυγραμμίζεται με τη βάση, με τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι ε, θα ήταν ιδανικό ένα κανονισμό που να είναι δεσμευτικό, να εφαρμόζεται σε όλου σε υψηλότερο βαθμό προστασία και με τι αυστηρότερε προδιαγραφέ. Το προτιμούμε αυτό από μια οδηγία φυσικά, αλλά θα δούμε αυτά και θα ολοκληρώσω εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κύριο Άλβαρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ να πιστεύω ότι όσο σημαντικό και να είναι το θέμα, μην νομίζουμε ότι θα πρέπει να ξαναφεύρουμε τον τροχό. Η αντίστοιχη οδηγία είναι πάρα πολύ καλή όπως είναι και όλα αυτά που λέει ο κύριος Φως υπάρχει μέσα το σύνολό τους, όλα αυτά που λέτε. Είναι το κλασικό δίκαιο από το 1995 και παγκόσμια είναι γνώμονα στο μεταξύ και κριτήριο, με εξαίρεση ίσω στις Αλλά υπάρχουν χώρες και στην Ασία που αυτό τον καιρό παίρνουν τη δική μας οδηγία και τη χρησιμοποιούν ω υπόδειγμα για να φτιάξουν δική τους νομοθεσία. Ποιο είναι το αποφασιστικό εδώ και δυστυχώ δεν αφορά την ίδια την οδηγία κανονισμό ότι θέλετε. Είναι η εφαρμοστικότητα, η εφαρμοσιμότητα, συγγνώμη. Ε, αυτό όμως δυστυχώς δεν είναι στο περιεχόμενο αυτού του φακέλου γιατί πολλές φορές είναι υπόθεση των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι αρκετά εφευρετική που για να ισχύσει το άρθρο 16 της θήκης Λισαβόνα. Αυτό που προτείνει η Σόφι Νετφέλτ για την επιβολή κυρώσεων ε, για την εφαρμογή. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα χρειαστεί να αντιπαρατεθούμε και με τα κράτη-μέλη γιατί σωστά ε, οι ποινικέ κυρώσει δεν είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Ε, στο περιβάλλον έχουμε καταφέρει όμως να το επιβάλλουμε αυτό, δεν ξέρω, ίσως και στην προστασία των δεδομένων. Κάτι άλλο τώρα που έχει αποφασιστική σημασία. Δεν είναι οι κλαδικές ρυθμίσεις, όσο σημαντικό ε, και αν είναι αυτό που συνέβη από το 1995 στο διαδίκτυο. Από το 95 τα έχουμε ρυθμίσει όμως για την ιδιωτική σφαίρα αυτό το privacy και να μην βάλουμε τώρα θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Τι δουλειά έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι προστασία των πολιτικών δεδομένων. Και αν ακριβώς λόγω της ψηφιοποίησης ε, ε, έχουν γίνει πρόοδοι και στο δημόσιο και στην ιδιωτική ζωή και στις εταιρείες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία, δηλαδή αυτή, η ασφάλεια των δεδομένων, αυτοί που συλλέγουν δεδομένα να ε, τα χειρίζονται με τον ασφαλή τρόπο. Πώς θα αποφύγουμε ζητήματα κατάχρησης ή ζητήματα να έχει ε, πρόσβαση κάποιος που δεν δικαιούται. Όλα αυτά είναι θέματα εφαρμογής για να μην φεύγουν από ε, της τράπεζας δεδομένων αυτά τα στοιχεία για αλότριους σκοπούς. Είναι και ο πρώτος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας. Γι' αυτό χρειάζεται αναθεώρηση η οδηγία 9546, γιατί δεν έχουμε πια αυτή τη ε, κατασκευή των πυλώνων, αυτό το αρχιτεκτόνιμα και χρειάζεται αλλαγή. Εγώ θέλω όντως να φέρει κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενιαία επίπεδα και κανένας να μην νομίζει ότι μπορούμε να ε, υποχωρήσουμε πίσω από τις ρυθμίσεις του 95. Τολμώ να το προβλέψω αυτό με το κοινοβούλιο, την παρούσα σύνθεση που έχει το κοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη νομίζω δεν πρόκειται να πάνε πίσω από το 95. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό να συνδείξουμε τον πρώτο με τον τρίτο ε, πυλώνα για την αστυνομική συνεργασία ε, και πώς μπορώ αυτά να τα συνδέσω με την εσωτερική αγορά. Γιατί και εγώ ανησυχώ για τις εταιρείε που φτιάχνουν προφίλ, που μας κατακλείζουν με διαφήμιση. Ε, αλλά αυτό είναι θέμα προστασίας και του καταναλωτού και να πούμε ναι ή όχι. Αλλά είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της προστασίας γιατί η ψηφιοποίηση δεν είναι κάτι που γίνεται ερήμην των ε, δημοσίων αρχών, γιατί υπάρχουν και κάποιες αρχές, κάποια ε, δημοτολόγια ας πούμε ή άλλου είδους αρχές που έχουν στοιχεία και προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να δούμε επίσης τα θέματα εθνικής ασφαλείας, πώς ορίζεται αυτή και είναι πάρα πολύ δύσκολο τις εξαιρέσεις να τις ελέγχουμε. Εάν ε, θέλει κανείς ε, να κάνει μια θαραλέα κίνηση να εξτάσει το θέμα των ορισμών και των ενιών. Τελειώνω, Πρόεδρε. Για τις διευθύνσεις IP δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά, τα έχουμε ρυθμίσει. Για την ε, οδηγία ή κανονισμός δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, θα πρέπει να είναι ένα πλαίσιο ευέλικτο, ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας και για το διασυνεριακό πρόβλημα, πώς μπορούμε να το λύσουμε ενδεχομένω. Όταν Έχουμε ε, προδιαγραφή ISO 9001 να φτιάξουμε και ένα ευρωπαϊκό σήμα, μια σφραγίδα για πιστοποίηση της ε, προστασίας των δεδομένων. Γιατί αυτό μπορεί να ελεγχθεί ε, εάν συμμορφώνεται ένα προϊόν και να φέρει αυτή τη σφραγίδα και να μπορεί να το αναγνωρίζει και ο καταναλωτής, ο πολίτης. Και τότε δεν με ενδιαφέρει αν η εταιρεία εδρεύει στον Πακού ή στο Παρίσι, εφόσον έχει αυτό το σήμα, αυτή τη σφραγίδα, ξέρω ότι έχει την πιστοποίηση, τη βούλα, ότι τηρεί ε, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δεν με νοιάζει αν είναι διασυνοριακή η, συναλλαγή. Αυτά. Και αυτό δεν είναι μόνο δικό μου. Τα έχουν σκεφτεί και οι Ιάπωνες, ξέρετε όλο αυτά. Ευχαριστώ και στην ανακοίνωση εν μέρη αυτό ε, συμπεριλαμβάνεται. Ο κύριος Άλμπρεχτ, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα και εσείς όσο γίνεται. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να μιλήσω αγγλικά. Δεν έχω πρόβλημα. <laughs> Ελληνικά βλέπει κάποιος. Ελληνικά κολλείομαι αυτή τη στιγμή. Ε, ε, στα αγγλικά τότε. Ο Άλεξ είπε πολλά ενδιαφέροντα σημεία και με κάλυψε, ήθελα να τα πω κι εγώ. Το σημαντικότερο είναι ότι η οδηγία 9546 είναι αφετηρία για όλη τη συζήτηση, βεβαίως. Τώρα ε, θα μεταφερθεί στην εποχή της Λισαβόνας, θα έχουμε νέο κανονισμό ή οδηγία, τι θα είναι αυτό, θα καλύπτει πρώτο και, δεύτερο, και τρίτο συγγνώμη, πυλώνα και ορισμένα πράγματα θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ε, πριν προχωρήσουμε. Μιλάμε πρώτα για οδηγία, για κανονισμό που δεν αφορά μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Αυτό ήταν ήδη σκοπός και πεδίο εφαρμογής πρώτης οδηγίας ε, του 1995. Αυτά δεν είναι εμπόδια. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της καταπολέμησης του εγκλήματος ή της τρομοκρατίας, ούτε και αυτό είναι εμπόδιο για την προστασία των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων είναι μια δυνατότητα και ένα πλαίσιο αποτελεσματικό για προστασία δεδομένων δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής, ε, διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων στην Ευρώπη και με τρίτες χώρες βέβαια ίσως, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των αρχών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποιες ρυθμίσεις και κανόνες το πρόβλημα της εφαρμογής ε, δεν εντοπίζεται μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εντός αυτής. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ποινές ή κυρώσεις αν υπάρξουν παραβιάσεις ε, ε, στη χρήση των δεδομένων. Το θέμα της πιστοποίησης, των μοντέλων πιστοποίησης επίσης θα πρέπει να το εξετάσουμε. Όλα αυτά όμως είναι δυνατά. Και είναι πολύ καλή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε λίγα σημεία. Για παράδειγμα, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμούμε τον κανονισμό από την οδηγία και ένα ευρύ περιεκτικό πλαίσιο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα συμφωνήσουμε ότι μια οδηγία ότι η οδηγία για, τα, την προστασία δεδομένων που είχαμε προηγουμένως είναι το σημείο αφετηρίας για μια βελτιωμένη προστασία και αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα πρέπει να διαμορφώσουμε τη θέση μας και να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποιες αρχές. Γενικώ έχουμε καλές αρχές στα μέτρα μας για την προστασία των δεδομένων. Αυτές τις αρχές θα πρέπει να τις κρατήσουμε και να επιβάλλουμε επιπλέον κανόνες για την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες τεχνολογίες στην εποχή του ίντερνετ με το cloud computing, το θέμα του profiling που είναι πολύ σημαντικό. Και αν μιλούμε για την εποχή του διαδικτύου, που καλύπτεται και από την οδηγία για την ιδιωτική σφαίρα, την ιδιωτική ζωή, αυτό το θέμα θα πρέπει να το καλύψουμε και στην οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Και θα πρέπει να μιλούμε για τη δυνατότητα της ανωνυμίας ή της παρουσίας με ψευδόνυμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για την ιδιωτική σφαίρα ή τον ενημερωτικό αυτό προσδιορισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που όλα είναι ε, αλληλένδετα. Γιατί μπορεί να μας φωτογραφίσει οποιοδήποτε και αυτός που μας τραβάει τη φωτογραφία μπορεί να μάθει τα πάντα για μας. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε αν αυτή η φωτογραφία συνδέεται άμεσα με μένα ως πρόσωπο ή απλώς με το ψευδόνυμο μου. Η κυρία Ένστιν είναι η τελευταία ομιλήτρια και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για μια σύντομη δευτερολογία. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Είναι γεγονός και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε ότι έχουμε οδηγία ε, για την προστασία των δεδομένων και μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα καινούριο, να αναπτύσσουμε νέες ιδέες. Να έχουμε ίδιες προδιαγραφές, εναρμόνιση της προστασίας, αυτό είναι σημαντικό, και ε, στην ποινική δίωξη και στην προστασία και πρόληψη του εγκλήματος. Πώς μπορούμε αυτό να το επιβάλλουμε σε όλους τους τομείς, δραστηριοτήτων και να έχουμε ένα ενιαίο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δυνατότητε έχουμε να δρούμε εκτό Ένωση με τα γνωστά προβλήματα. Η προστασία των δεδομένων θα πρέπει καταρχήν να είναι δεδομένη για όλου. Θα πρέπει να το έχουμε και στο μυαλό μα αυτό σαφέ. Ίσως χρειαστεί να σκεφτούμε περισσότερο ειδικού τομεί, όπω τι γίνεται με την προστασία των εργαζομένων, των, των δεδομένων των εργαζομένων. Δεν λέω ότι θα πρέπει να το γράψουμε εδώ έτσι ρητά, αλλά να το σκεφτούμε, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες εκεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η συζήτηση για την παρακολούθηση της εφαρμογής. Και τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης ε, της συνθήκης. Έχουμε νομικά μέσα στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ένα άλλο ακόμα είναι τι χρειάζονται πραγματικά οι πολίτες ε, ως προστασία των δεδομένων τους, των προσωπικών τους δεδομένων. Να υπάρχει πραγματική διαφάνεια, όχι στα λόγια. Εύκολη πρόσφαση, ε, νομική βοήθεια, προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια και πάνω να είμαστε και φιδωλοί με τη διάδοση των προσωπικών μας δεδομένων. Κάτι άλλο που θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το πω είναι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εποπτών των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Να είναι πάντα ε, σίγουρη και ενισχυμένη η ανεξαρτησία αυτών των αρχών και να έχουν και τις ε, αντίστοιχες αρμοδιότητες. Και ένα τελευταίο. Δεν μου αρέσει αυτό που λέμε για τις ελάχιστες προδιαγραφές στην προστασία των δεδομένων. Γιατί ελάχιστες, όσο γίνεται ευρύτερε προδιαγραφές να έχουμε να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό και τι θέλουμε πραγματικά. Και οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φως, σύντομα σας παρακαλώ. Είδατε ότι γενικά σας υποστηρίζουν οι συνάδελφοι, αλλά παρακαλώ έχετε το λόγο για να κρυώσετε. Ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τόσο σύντομα σε όλα αυτά τα θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Φαίνεται σας τρόμαξα όταν μίλησα για μια νέα ματιά, μια φρέσκια ματιά. Δεν είπα να καταργήσουμε την οδηγία εντελώ. Φυσικά και είναι αφετήρια των σκέψεών μας και του προβληματισμού. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε όλα αυτά στα καινούργια δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Βεβαίως, Μπορεί κάποιος να έχει ακτιμήσεις, αξιολογήσεις για το αποτέλεσμα της οδηγίας, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτά. Ορισμένα πράγματα που αναφέρατε, δεν ξέρω αν ήταν κριτική σε αυτά που είπα εγώ, πάντως ορισμένα από αυτά που άκουσα, ε, είναι για μένα δεδομένα. Είτε έχω επιβεβαιώσει, είτε είχα πει κι εγώ. Δεν ξέρω. Ε, Μηπω δεν ήμουν αρκετά σαφή επειδή είπα τόσα πολλά. Και το τελευταίο για τις ελάχιστες προδιαγραφές. Εγώ δεν θέλω να έχω ελάχιστες ή μέγιστε προδιαγραφές. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας. Παντού το ίδιο. Και σε υψηλό επίπεδο όμως. Ε, δεν ξέρω πώς θα τα πούμε αυτά τα στάνταρ ελάχιστες προδιαγραφές ή όχι. Να ενισχύει παντού το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θέλω εγώ και μάλιστα σε αρκετό υψηλό βαθμό. Γιατί αυτό που ήδη ισχύει είναι αρκετά υψηλό και δεν θέλουμε να ε, πέσουμε σε επίπεδα κατώτερα το 95 να το βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου είπατε. Θα τα λάβω υπόψη μου και θα τα συμπεριλάβω και στο σχέδιο της έκθεσής μου και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το επίπεδο για να ε, προκύψει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο σύγχρονο, λογικό και ωραίο. Ευχαριστώ. Ναι, αναγνώριση. Υπάρχει και ήταν ορατή η υποστήριξη όλων των συναδέλφων. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Αυτή της απογευματινής τη Πέμπτης θα ήθελα να καλέσω του δύο γενικού διευθυντές στο Προεδρείο. And, uh, this, this point is, uh, the, um, Σήμερα θα έχουμε την πρώτη συζήτηση για τα θέματα που ενδιαφέρουν uh, την Επιτροπή μας στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013. Όπω ξέρετε και η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ ασχολείται με τα θέματα αυτά του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε κοντά μα δύο γενικού διευθυντέ από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που θα μα εκθέσουν τι απόψει του για τις εξελίξεις και θα μα μιλήσουν για, τη, για το πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Η, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στα πλαίσια του 3 είναι γιατί είναι τη, για τους πρόσφυγες και τα σχετικά κονδύλια, τη μετανάστευση κτλ. Και, έχουμε το γενικό πρόγραμμα για τη διασφάλιση των πολιτικών ελευθεριών και επίσης είναι αρμόδια για τους οργανισμούς Frontex, ES, SEPOL, Europol και, το μελλοντικό οργανισμό καθώς και την ε, ανάπτυξη του συστήματος Eurodac. Έχουμε συζητήσει πολλά πολλά, πολλά εξ τα θέματα. Και η Γενική Διάθεση Δικαιοσύνη ασχολείται με το πρόγραμμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια, ε, ποινική δικαιοσύνη, ε, ναρκωτικά, θέματα αποτοξίνωσης, ε, εθισμού στα ναρκωτικά κτλ. Και μετά την εισαγωγή θα έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μανσερβίση το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων και κατόπιν στην κυρία Λεμπάγη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κάποιες σκέψεις για το μέλλον, βασικές προτάσεις. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για πιο λεπτομεριακές αναλύσεις. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, ο μηχανισμός εσωτερικών υποθέσεων είναι 0,77% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού, 6,4 δις για την περίοδο 2007-2013. Αυτό καλύπτει τα προγράμματα, τους οργανισμούς και τα μεγάλα συστήματα IT, πληροφορικής και τεχνολογιών. 4 δισεκατομμύρια αφορούν τα γενικά προγράμματα ε, αλληλεγγύη και διαχείριση της μετανάστευσης, που ε, προβλέπονται από τα τέσσερα ταμεία προσφύγων, ένταξης, ε, εξωτερικών συνόρων και επαναπατρισμού και έχουμε 100 εκατομμύρια για το Γενικό Πρόγραμμα Ασφάλειας και Πολιτικών Ελευθεριών που εμπίπτει στην, κεντρική διαχείριση, ενώ οι οργανισμοί καλύπτονται κατά 18% του προϋπολογισμού, από το 18% του προϋπολογισμού, Europol, Sepol, Frontex, ε, Κέντρο Παρακολούθηση για τα Ναρκωτικά, η ΆΣΟ και η ο Μελλοντικό Οργανισμό για τι Τεχνολογίε τη Πληροφορική, που θα καλύψει το ΣΥΣ, το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν και άλλου μηχανισμού μάλλον. Και σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων, θα ήθελα να πω ότι είναι κάπω παράδοξο ο τρόπο. Είναι ένα περίεργο παράδειγμα backloading ξεκινούμε από χαμηλά ποσά και στο 2013 έχουμε μεγάλη αύξηση. Επίσης έχουμε αιτήσει αύξηση 15%. Αυτό να το λάβουμε υπόψη. Για δύο λόγους γίνεται η αύξηση αυτή. Καταρχήν για να επιτρέψουμε τη διαδικασία τα κράτη-μέλη να εκταμιεύσουν και να βελτιώσουν το ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων. Και επίσης έχουμε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στους τομείς αυτούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί θα αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας ε, για το σχεδιασμό των ποσών και το ύψο των ποσών για την επόμενη περίοδο, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά είναι πάνω κάτω τα ποσά, τα ξέρετε φαντάζομαι. Δεύτερον τώρα, ποιε είναι οι αδυναμίε του ισχύοντο συστήματο. Θα έλεγα κατά βάση ότι έχουμε δύο είδη προβλημάτων και αδυναμιών. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε σήμερα να δράσουμε αμέσως για να ανταποκριθούμε σε μια κρίση, για να βοηθήσουμε κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μια κρίση ή να βοηθήσουμε εταίρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή να λάβουμε πρωτοβουλία και να βοηθήσουμε κάποιους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Για παράδειγμα, επαναπατρισμό των ε, κατοίκων Ερθρέας ε, και Σομαλίας που βρίσκονται μεταξύ Λιβύης ε, Αιγύπτου και την Ισία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, γιατί είναι τόσο γραφειοκρατικό και ε, βραδικίνητο το σύστημα που ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια θέματα. Δεύτερον, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε μικτές ε, ε, ομάδες ερεύνης. Κάτι που είναι σημαντικό για την εξάρθρωση διεθνών κυκλωμάτων εγκλήματος. σε ό,τι αφορά τα συνοδευτικά μέτρα. Και εκεί έχουμε προβλήματα για τα συμπληρωματικά ποσά. Και εκεί υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα. Και τέλος, δεν μπορούμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας απέναντι στις τρίτες χώρες. Γιατί πολύ συχνά όταν έχουμε εντολή συμφωνία παρισδοχή ακόμη και συμφωνία εταιρικής σχέσης, δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας και να εξασφαλίσουμε ε, την αποδοχή και εφαρμογή μιας συμφωνίας επανεισδοχής και από τη στιγμή που επαναπατριστούν οι ενδιαφερόμενοι να τύχουν σωστής ε, αντιμετώπισης από τη χώρα προέλευσής τους. Ούτε μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε δράσεις που θέλουν να ενισχύσουν το δυναμικό της χώρας για την καλύτερη διαχείριση των σύνορων. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ή μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά α, με κάποιους α, παράλληλους δρόμους που όμως ε, εξαρτώνται από άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μηχανισμούς. Αυτές ε, είναι αδυναμίες του μηχανισμού παράδοσης. Επίσης, ο μηχανισμός αυτός έχει τέτοια χαρακτηριστικά που αντί να αναλαμβάνει τους κινδύνους της μετανάστευσης και τον ε, δεχόμενο κίνδυνο μιας ε, χώρας που αντιμετωπίζει μια κρίση ή το θέμα της κατανομής των κονδυλίων για τα εξωτερικά σύνορα, όλοι οι μηχανισμοί είναι μαθηματικοί και αντικειμενικοί, αλλά αντί να κοιτάς στο μέλλον, κοιτάς στο παρελθόν. Οπότε, πολύ συχνά, ένα κράτος που σε μια δεδομένη χρονιά χάρη της ε, επένδυσης είχε καλή διαχείριση, όχι μόνο δεν θα επιβραβευθεί, αλλά θα πληγεί κιόλα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τι συνέβη στο παρελθόν και όχι το πώς συνέβη και, και βλέπουμε ποιος είναι ο αντικειμενικός κίνδυνος για το μέλλον. Αυτό είναι προβληματικό και για τη διαχείριση των συνόρων και ισχύει και για την αντιμετώπιση των προσφύγων. Όλα αυτά τα κονδύλια αντί να στρέφονται προς το μέλλον, είναι στραμμένα προς το παρελθόν. Και αντί να προβλέπουμε τα γεγονότα, ουσιαστικά είμαστε οραγοί και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Η ταξινόμηση επίσης είναι πολύ παραδοσιακή, παροχημένη σχεδόν και κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 100 προγράμματα και προγράμματα εργασίας. Κάθε χρόνο δηλαδή, κάθε ταμείο εξετάζει το πολιετές πλαίσιο που υπευλήθη στην αρχή του έτους και κάθε χρόνο έχουμε και τα ετήσια προγράμματα που είναι σχεδόν 27 ή αν όχι 27, σχεδόν 27. Συνήθως έχουμε 27 επί 4 και αυτό σημαίνει προγραμματισμό, παρακολούθηση, έλεγχο και κλείσιμο, καθάριση. Φανταστείτε τι προσωπικό χρειάζεται και τι ενέργεια μόνο για τη διαχείριση του περιορισμού του κινδύνου σε τη φορά τη χρηματοπιστωτική διαχείριση. Και αν πρέπει να επέβουμε σε αυτόν τον οργανισμό και να εφαρμόσουμε και κάποια ελαστικότητα, τότε έχουμε παραλύσει τελείω. Αυτή είναι μια δεύτερη σοβαρή αδυναμία. Επίσης, πρέπει να το δείτε με τα μάτια σα και να το πιστέψετε. Κάθε ταμείο έχει τη δική του νομική βάση, του τέστην. Υπάρχει κατακόρυφος διαχωρισμός και πολύ συχνά έχουμε επικαλύψεις. Αντί να εφαρμόζουμε, αντί να θεσπίζουμε στόχους, ουσιαστικά εφαρμόζουμε μέσα που μερικές φορές είναι κατάλληλα για την υλοποίηση των στόχων μας. Τώρα, αυτά αυτές είναι δυναμίες και από ουσιαστική αλλά και από διαδικαστική άποψη. Τώρα, ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ταμείων που θα πρέπει να προβληθεί, να προβληθεί και να συζητηθεί. Θα σας δώσω και πάλι μερικά παραδείγματα γενικά και μετά αν θέλετε επισερχόμαστε και σε λεπτομέρειες. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Είχαμε πρόσφατες συζητήσεις για την ε, διεύρυνση, επέκταση του χώρου Σέγγεν. Και εδώ είναι θέμα πώς θα βοηθήσουμε διαρθρωτικά κάποια κράτη που έχουν διοικητικέ αδυναμίες, αλλά επειδή έχουν εξωτερικά σύνορα τη Ένωση είναι επιφορτισμένα με την προστασία ολόκληρη τη Ένωση. Αν ε, εγκριθεί η νομική βάση για το σύστημα αξιολόγηση έγκεν, θα θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη και να διαθέτουμε και σχετικά κονδύλια να το κάνουμε φυσικά. Επίση, να αλλάξουμε την προσέγγιση για τη διαχείριση των σύνορων. Και όχι απλώ να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα τα κράτη που έχουν τα εξωτερικά σύνορα υποχρεούνται να κάνουν κάτι. Χρειαζόμαστε ένα είδους που είναι προ όφελο ολόκληρη τη κοινότητα. Γιατί οι πολίτες θα έχουν εμπιστοσύνη στα εξωτερικά σύνορα αν η διαχείριση γίνεται με εναρμονισμένο τρόπο, με βάση ποιοτικέ προδιαγραφές, με αξιοπιστία των αρμοδίων αρχών. Δεν θα υψέλθω τώρα στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ακριτοφυλακή. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι χώρες εξυπηρετούν το συνολικό συμφέρον και δεν είναι μόνες τους, όχι μόνο το δικό τους. Οπότε, πέραν της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την υπηρεσία με τη χρήση των διαφόρων οργανισμών, που δεν θα είναι μόνο οι σανίδα σωτηρίας, αλλά θα προσφέρουν και διαρθρωτική υποστήριξη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στην Νότιο ε, στη Νότια Λιθουανία. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, γιατί έχουμε ανθρώπου που χρειάζονται προστασία, έχουμε χώρε που χρειάζονται προστασία και έχουμε και ένα περιφερειακό σύστημα προστασία, ώστε άνθρωποι που χρήζουν διεθνού προστασία να την λάβουν. Υπάρχει και το πρόβλημα τη επανεγκατάσταση. Δεν είναι δίκαιο ο καταμερισμό του άχθου στην Ευρώπη αλλά δεν έχουμε και μέρο, με, μέσα στη διάθεσή μας υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια μέσα και μηχανισμούς για να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η νέα πραγματικότητα του διασυνοριακού εγκλήματος ή του κυβερνοεγκλήματος ή των τρομοκρατικών απειλών οι προκλήσει αυτές είναι τόσο τεράστιες που δυστυχώ δεν έχουμε αρκετά οικονομικά μέσα για να ανταπεξέλθουμε. Χρειαζόμαστε και περισσότερες γνώσεις και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Επίση, ό,τι αφορά τι εξωτερικές δράσεις, το είπα ότι χρησιμοποιούμε κάποια μέσα που έχουν προσδιοριστεί περισσότερο για λόγους ανάπτυξης για έξι χρόνια ήμουν Γενικός Διευθυντής σε θέματα ανάπτυξης και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτά τα ε, μέσα που είχαν αναπτυξιακό στόχο για τις χώρες δικαιούχους τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνουν αυτές οι χώρες ε, αξιόπιστοι εταίροι και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει μια μεγάλη διχοτόμηση εδώ. Το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη έκθεση. Και αν η πολιτική μας επανεισδοχής ε, δεν συνοδευτεί από τα απαραίτητα οικονομικά μέσα θα είναι μια αποτυχία. Και δεν έχουμε μόνο τα θέματα επανεισδοχής, έχουμε τα θέματα της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα. Αν δεν έχουμε ε, μέσα που θα είναι και εμόχλευση για μεταρρυθμίσεις, τότε δεν θα επιτύχουν οι πολιτικέ μα Και αν δεν έχουμε κονδύλια ώστε όσοι επιστρέφουν στι πατρίδε του να τύχουν δική αντιμετώπιση, να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, τότε αν δεν τα εξασφαλίσουν όλα αυτά είναι κενό γράμμα οι πολιτικέ μα. Σα έδωσα λίγα παραδείγματα για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά και τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να υλοποιήσουμε τι προτεραιότητέ μα. Θέλουμε και μια πλούστευση του όλου συστήματος. Σας μίλησα για τους οργανισμούς, για τα κονδύλια, τα ταμεία που έχουμε. Θα πρέπει καταρχήν να μειώσουμε τον αριθμό των ταμείων, να τα, να τα συγκεράσουμε σε δύο. Το ένα ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση και το, άλλο, το δεύτερο ταμείο για διαχείριση συνόρων και ασφάλεια. Να μειώσουμε τον αριθμό των ταμείων, να περιορίσουμε τον κατακαιρματισμό και να κάνουμε τα ταμεία πιο φιλικά προς το χρήστη. Επίσης, να σταματήσουμε αυτό τον επιβλαβή συνδυασμό μεταξύ των, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των ετήσιων προγραμμάτων. Γιατί αυτό επιτείνει τη γραφειοκρατία. Καλό θα είναι να έχουμε έναν πολιετή προγραμματισμό που θα, θα μεταφράζεται σε αιτήσει δράση. Αλλά να μην έχουμε κάθε χρόνο νέα διαπραγμάτευση. Γιατί έχουμε πάνω από 100 προγράμματα. Δεν μπορούμε ετησίω να τα εξετάζουμε. Τρίτο ζήτημα της απλούστευσης. Συστηματική χρήση της ε, κοινή διαχείρισης. Μεταρρυθμισμένης όμως κοινή διαχείρισης. Γιατί η κοινή διαχείριση σημαίνει κατανομή μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων. Και κάθε χρόνο βλέπουμε τι συμβαίνει και κάνουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Πάντως, με βάση απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση τη κοινή διαχείριση, θέλουμε η κοινή διαχείριση να γίνει ένα συμβολέου για, για την υλοποίηση των στόχων. Αντί να μοιράζουμε δηλαδή χρήματα και να βλέπουμε εκ των υστέρων τι συμβαίνει, να προσδιορίζουμε εκ των προτέρων με τη βοήθεια των κρατών μελών και στη συνεργασία μαζί του, ποιοι στόχοι θα επιδιωχθούν από κάθε κράτο που δεν είναι κατά αναγκή ίδιοι. Και μετά με δείκτε να έχουμε και πιο διαφανή και πιο συγκροτημένο διάλογο με τα κράτη-μέλη και στο τέλος να καταμετρήσουμε αν υλοποιήθηκαν ή όχι οι στόχοι. Κοινή διαχείριση μεν, αλλά μεταρρυθμισμένη κοινή διαχείριση για να υλοποιήσουμε τους στόχους. Αυτό εξετάζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την εμπειρία που είχαμε από το γενικό τρόπο διαχείρισης, της κοινής διαχείρισης. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις, την έκτακτη, τις έκτακτες, κατεπίκουσες περιπτώσεις. Αν είχαμε και εμεί τέτοια κονδύλια περισσότερα, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και περιπτώσεις έκτακτη ανάγκη ε, και να βοηθήσουμε χώρες που αντιμετωπίζουν κάποια κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη είναι πολύ περιορισμένη πολλές φορές έχουμε απρόβλεπτες, ε, απρόβλεπτους κινδύνους, μετανάστευση, τρομοκρατικές απειλές ή ανάγκη διεθνούς προστασίας. Μέχρι στιγμής τέτοιες δυνατότητες δεν έχουμε. Και τέλος, ο ρόλος στον οργανισμό που εντάσσεται σε αυτό το προβληματισμό της απλούστευσης του όλου οικοδομήματος. Αυτό που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή ο ρολος των οργανισμο που εντασσεται σε αυτο το προβληματισμο της είναι να χρησιμοποιήσει τους οργανισμούς σε ένα πιο εύληπτο για τον κόσμο πλαίσιο και πιο κατανοητό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη. Και οι οργανισμοί να αποτελέσουν τμήμα της εργαλειοθήκης της Ένωσης και να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της. Να, γίνουν οι οργανισμοί, να αποκτήσουν οι οργανισμοί και ένα εκτελεστικό ρόλο. Βέβαια είναι ρυθμιστικοί όλοι αυτοί οι οργανισμοί και δεν το λέω από τεχνική άποψη το θέμα το εκτελεστικό, αλλά στο πλαίσιο ενός προγράμματος που υποστηρίζει τις συστηματικές προσπάθειες των κρατών μελών για τη διαχείριση των συνόρων, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη Frontex για μόνιμη τεχνική αρρωγή προς τα κράτη-μέλη που χρειάζονται και τεχνογνωσία και υποστήριξη, αλλά και αλλαγή των ποιοτικών προδιαγραφών. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτού του οργανισμού και κατά ανάγκη με αύξηση του προπολογισμού του, αλλά να του χρησιμοποιήσουμε για συγκεκριμένου σκοπού με βάση ad hoc ε, χρηματοοικονομικά προγράμματα. Έτσι θα αυξήσουμε και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των οργανισμών και θα προσδιορίσουμε και στόχους σε πολιτικό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταστήσουμε τους οργανισμούς ως εκτελεστικούς, θα τους καταστήσουμε εκτελεστικούς βραχίονες κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που δεν είναι αμυγός εκτελεστικά όργανα. Αλλά μπορούμε να έχουμε ένα είδος action on demand, κατά παραγγελία δράση από τους οργανισμούς, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ήμουν υποχρεωμένος ναι. να μείνω σε γενικές παρατηρήσεις και να τηρήσω και το χρόνο. Πάντως αυτές ήταν οι αδρές γραμμές Τη ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι έχουμε, τι χωλαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, πλησιάζουμε προς το τέλος ε, του προηγούμενου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Οπότε έχουμε ήδη μπει σε μια ε, ταχύτητα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Παρακαλώ την κυρία Λεμπάη να πάρει το λόγο και μετά μπορούμε να κάνουμε ερωτήσει ή σχόλια και εμεί. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά δικαιοσύνη, ο προπολογισμό είναι μικρό, Ένα δισεκατομμύριο έχουμε για την τρέχουσα 7 περίοδο. Είναι ένα δισεκατό του συνόλου του προπολογισμού της Ένωσης. Δεν είναι και τεράστιο το ποσό. Αλλά από αυτό το 1 δις 36% πηγαίνει ε, στους οργανισμούς, γνωρίζετε τους οργανισμούς. Είναι ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, για την Ισότητα των Φύλων, Eurojust κτλ. Και βεβαίως ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ποσοστό του προπολογισμού που πηγαίνει εκεί και κατά τα άλλα έχουμε πέντε προγράμματα τα οποία έχουμε αναπτύξει με την πάροδο των ετών, με τις διάφορες πολιτικές που ε, λαμβάνουν χώρα και υλοποιούνται. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι ε, κοιτάξαμε τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούν αυτά τα προγράμματα, τα έχουμε αξιολογήσει και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής δεν μας εκπλήσει καθόλου. Έχει αποδειχθεί ότι τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά εκτός αυτού είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα είναι ε, ανα, περίπτωση, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ε, της κάθε περίπτωση είναι μικρό πρόγραμμα με βαριά γραφειοκρατία, με βαριά ε, διοίκηση και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών θεωρεί ότι υπάρχει χώρος ε, βελτίωση αυτών των προγραμμάτων. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν στο μέλλον γι' αυτό και ε, πάρα πολύ στις γραμμές που ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνολική θεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Είδαμε την προστιθέμενη αξία την υποστήριξη των βασικών προτεραιοτήτων πολιτικής, πολύ σημαντικό και αυτό. Και επίσης ε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα αποτελέσματα, εκεί προσανατολιζόμαστε. Και ε, ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να δούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε το πραγματικό αντίκτυπο ε, της βοήθειας που παρέχεται και ε, αυτό μας απασχολεί και μας προβληματίζει, όπως και η ουσία. Τι χρειάζεται δηλαδή ε, η δικαιοσύνη τα επόμενα χρόνια. Uh, και ε, σε θέματα δικαιοσύνης λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι η εφαρμογή των πολιτικών. Πρόσφατα έχουμε ε, αναπτύξει και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να αναπτύσσουμε ένα ολόκληρο σύνολο ε, νομοθετικών μέσων. Για τη δικαιοσύνη όμως δεν αρκεί να εγκρίνεις κάποια μέσα, χρειάζεται και πραγματική εφαρμογή και να έχεις τα στοιχεία εκείνα που θα διασφαλίσουν την πραγματική εφαρμογή των νομικών μέσων. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να αναπτυχθούν. Πρώτον, ε, κατάρτιση και είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος της Στοχόλμης που μας καλεί να εκπαιδεύσουμε τους μισούς νομιμομαθείς στην Ευρώπη που είναι 600.000 εάν δεν εκπαιδεύεις ε, δικαστές, αν δεν εκπαιδεύεις δικηγόρους στην ε, εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για το μέλλον πολύ μεγάλη προτεραιότητα είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών. Προηγουμένως συζητούσα την προστασία των δεδομένων, αλλά εκεί ας πούμε θα χρειαστεί οπωσδήποτε ε, στα πλαίσια της νέας μορφής σχεδιασμού θα χρειαστεί, λέω, πολύ μεγαλύτερη συνεργασία, πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών και εποπτών προστασίας προσωπικών δεδομένων με αλληλοκατανόηση και των αναγκών του καθενός έτσι ώστε οι ερμηνείες που δίδονται να είναι ίδιες. Αυτό είναι ένα και μόνο παράδειγμα το οποίο όμως σας δίνει μια ιδέα για τη σημασία που μπορεί να έχει η εκπαίδευση και κατάρτιση. Άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό επίσης είναι η ανάπτυξη ε, εργαλείων ε, ηλεκτρονικών. Πρόσφατα δημιουργήσαμε το e-Justice, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Δεν είναι άλλη μία ιστοσελίδα. Είναι πάρα πολύ λειτουργική αυτή η ιστοσελίδα, ο ιστότοπος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαστικές αρχές θα μπορούν να συνεργάζονται, να γνωρίζουν το νομικό καθεστώς και το, το νομικό παρελθόν μάλλον, ε, το μητρό ενός υπόπτου και είναι κομβικό αυτό για τη συνεργασία των διαφόρων νομικών μέσων που έχουμε ας πούμε, στο οικογενειακό δίκαιο. Ε, κρίσιμα, κρίσιμα αυτά τα θέματα πάρα πολύ και σημαντικότατα. Ε, ένα άλλο στοιχείο είναι η διασυνοριακή συνεργασία. Στη δικαιοσύνη αυτό βεβαίως ε, είναι ένα σημείο κλειδί και ε, δικαιοσύνη με την ευρία έννοια έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εξαφάνιση παιδιών. Όταν θα πρέπει πολύ γρήγορα να αντιδρούμε για να βρίσκονται τα παιδιά στα πρώιμα στάδια της εξαφάνισης. Ε, ένα άλλο στοιχείο εξίσου σημαντικό. Καλό είναι να αναπτύσσουμε τα δικαιώματα, αλλά οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Τι να το κάνεις το δικαίωμά σου και πώς να απαιτήσει να ε, εφαρμοστεί και να το διεκδικήσεις αν δεν ξέρεις καν ότι το έχεις αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή και αυτό μας απασχολεί στον επαναπροσανατολισμό ε, των προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση και Όλα αυτά είναι προκαταρκτικές βεβαίως σκέψεις και δράσεις και μετά έχουμε όλο το θέμα τη μεταφορά στην πράξη. Είναι πέντε τα προγράμματα, θέλουμε πολύ να τα απλουστεύσουμε και να υπάρχει τελικά ίσω ένα πρόγραμμα που να τα συνδυάζει, να τα συνενώνει όλα αυτά σε μια ε, ενότητα. Όλε αυτέ τι θεματικέ προτεραιότητε που έχουμε στα θεμελιώδη δικαιώματα, είτε στην ποινική δικαιοσύνη, είτε στην αστική δικαιοσύνη. Και να είναι και πιο εύκολη η εκτέλεσή τους στην πράξη για εκείνους που είναι δικαιούχοι των ε, χρημάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό και ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε αυτές τις πολιτικές ε, τι χρήματα δίνουμε αλλά και πού ακριβώς θα ε, πηγαίνουν αυτά τα χρήματα που μας δίνει η Δημοσιονομική Αρχή. Ευχαριστώ. Τώρα μιλούμε για ένα μικρό μόνο κλάσμα του συνολικού ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένας τομέας που καλπάζει στην ανάπτυξή του και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι στο μέλλον ότι θα έχουμε αρκετούς οικονομικούς πόρους για να καλύψουμε όλα τα προγράμματα και τις ε, αυξανόμενες ε, ανάγκες. Είδαμε τώρα και την πρόσφατη κρίση στην νότια όχθη της Μεσογείου και αυτό είναι ανησυχητικό ε, σημάδι. Χρειάζεται επιτάχυνση και ευελιξία σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχω τώρα τους εξής συναδέλφους. Αλβάρο, Κέλλερ και λοιποί. Πρώτος ο κύριος Αλβάρο και μετά βλέπουμε. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερα ε, τους δύο ε, προσκεκλημένους μας για την εκτενέστατη παρουσίαση. Ε, βασικά μιλάμε για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και καλό είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, που είμαι επίσης μέλος εκεί, συζήτησε σήμερα αυτά τα θέματα. Βέβαια, τα λέει εδώ, αλλά όχι εκτενώς η έκθεση. Καμιά φορά και οι ίδιοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τον προπολογισμό ε, δεν έχουν επίγνωση αυτών των θεμάτων, υποτιμούν τα θέματα. Ξέρετε, είναι η έκθεση Γκαρίγκα που καλύπτει το πολιετές πλαίσιο όλο τον προεπολογισμό της Ένωσης. Ε, μπορεί να, περιορισμένα μόνο να φέρετε στα δικά σας θέματα, αλλά χάρηκα που τα άκουσα γιατί ε, είχα τη χαρά να το συζητήσω και με την Επίτροπο. Ήρθε και στο Στρασβούργο στην Επιτροπή Σούρε και πρότησε να έχουμε δύο ταμεία. Ένα για την ασφάλεια, ένα για τη μετανάστευση που το θεωρώ πολύ λογικό και σκόπιμο. Τι θα γίνει ε, με τη πολιτική γειτονία, δεν θα ήταν καλό να μπει ε, και στον τίτλο γιατί ουσιαστικά αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Πολλά προγράμματα το πηγαίνουν χέρι-χέρι, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη Βόρεια Αφρική. Είναι πολλά από τα προγράμματα της γειτονίας που υλοποιούνται εκεί. Θα ενδεχομένως να είχε νόημα να το εντάξουμε και αυτό ε, στο χαρτοφυλάκιο της εσωτερικής πολιτικής, γιατί η πολιτική γειτονίας πάντα επηρεάζει τα τεκτενόμενα εντός της ενώσεως. Δεν είναι πάντα θέματα ασύλου ή μετανάστευση. Συνεργαζόμαστε και με τη Ρωσία και με τη Λιθουανία τώρα για τα δίκτυα και έχουμε και ροές εργαζομένων, ανταλλαγέ. Δεν ξέρω, ίσως θα είχε νόημα να μπει και αυτό στη εσωτερικά και δικαιοσύνη. Τώρα το έχουμε στο σημείο 3. Δεν το αναφέρετε, δεν περίμενα να το κάνετε ε, εμείς θα το καταπολεμήσουμε. Τώρα προτείνεται με ΑΙ να υπάρχει ένας τίτλος ε, δύο ε, που, να ονομάζεται ιδιότητα του πολίτη, citizenship. Εκεί θα έχει διάφορα πράγματα μέσα γιατί είναι νεολαία και ε, διάφορα άλλα. Ο παλιός τίτλος 3. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσατε να μας το σχολιάσετε οι συνάδελφοι του Λαϊκού Κόμματος Εάν συμφωνείτε να επηρεάσετε τον κύριο Γκαρίγκα κάπως, γιατί στο μέλλον δεν έχει νόημα να έχουμε ένα τίτλο πολίτες, η ιδιότητα του πολίτη και να είναι ένα τσουβάλι που να τα ρίχνουμε όλα μέσα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική η νεολαία, η επικοινωνία, αλλά είναι άλλη ιστορία τα, ε, θέματα ε, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Δεν μπορούν να μπουν όλα μαζί. Εγώ σας υποστηρίζω και ελπίζω να καταλήξουμε και στην έκθεση σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Τώρα αυτό το καιρό κάνουμε τροπολογίες και εγώ και το γραφείο μου με χαρά να δεχτούμε και προτάσεις και σχόλια για την έκθεση ΣΟΥΡΕ και ε, από πλευρά τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά μην ξεχνάτε ότι μα χρειάζονται και τα κράτη-μέλη. Και αν διαφωνούν τα κράτη-μέλη, το πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο μπορεί να πάει σε άλλη κατεύθυνση, δημοσιονομικό καλύτερα, ο τίτλος να παραμείνει όπως έχει τώρα και όχι μια σούπα ε, για τον πολίτη γενικώ. Και με την πολιτική γειτονία στο τίτλο 3 που ουσιαστικά είναι σήμερα δικό σας, γιατί είναι πολλές οι συνέργειες εκεί και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να κάνουμε και οικονομίες στο κόστος, το διοικητικό και το γραφειοκρατικό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ. Άκουσα και εγώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους δύο γενικούς διευθυντές και έχω μερικές απορίες σε ό,τι αφορά τους τρόπους κοινή διαχείρισης. Στην Επιτροπή ΣΟΥΡ η Επιτροπή μας είπε ότι θέλει να επεκτείνει τη χρήση της κοινή διαχείρισης και είπατε θέλετε να τη μεταρρυθμίσετε και όλα. Φαντάζομαι πάνε μαζί αυτά. Σε ποιους τομείς θέλετε κοινή μεταχείριση, κοινή διαχείριση, συγγνώμη, αφορά και το εξωτερικό σκέλος αυτή η κοινή διαχείριση. Για ποιους τομείς τη σκέφτεστε. Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες να έχουμε ένα ταμείο για την εξωτερική διάσταση στο κεφάλαιο 3, στη Γενική Διάθεση Εσωτερικών Υποθέσεων. Γιατί είπατε ότι δεν έχετε κονδύλια για να μπορείτε να πρόσπισετε το κοινοτικό συμφέρον. Χαίρομαι που το επισημάνατε. Γιατί πολλές φορές ε, προσπαθεί η να μας πείσει ότι πρόκειται για το συμφέρον των ε, χωρών, των αναπτυσσομένων χωρών. Αλλά μερικές φορές οι δράσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εκρίζωση της φτώχειας. Και πώς θέλετε ακριβώς να το διαρθρώσετε. Δημοσιονομική γραμμή στο κεφάλαιο 3. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η γραμμή. θεματικά προγράμματα ε, όπως μετανάστευση στα πλαίσια του DCI. Ε, ή το μη αναπτυξιακό σκέλος θα Μιλήσατε και για τις συμφωνίες επανεισδοχής που χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από τα θεματικά προγράμματα. Τι θα γίνει, δεν χρειάζεται πια αυτό. Και ποια είναι η στρατηγική σας για την ε, χρησιμοποίηση των κονδύλιων της εξωτερικής διάστασης. Δεδομένων των εξελίξεων στη Βόρεια Αφρική, είδαμε ότι μέχρι στιγμή τα θεματικά προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν για συνεργασία, για, συνορι... για συνοριοφύλακε κτλ. Τι συμπεράσματα, σε τι συμπεράσματα κατάληξαμε τις επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική. Και τέλος, το σύστημα των δύο πυλώνων. Ένα μεγάλο ταμείο για την ε, μετανάστευση και ένα άλλο ταμείο για την ασφάλεια στα σύνορα ποιο είναι το πλεονέκτημα α, τη συγχώνευση σε δύο μόνο ταμεία, γιατί στο Ταμείο Μετανάστευση θα, είχα, περιληφθεί το Ταμείο των Προσφύγων, του Επαναπατρισμού ή της Επανεισδοχής. Δεν είναι ίδιες όμως οι αρμοδιότητες. Με ποια επιχειρήματα στηρίζεται αυτή την πρόταση για συγχώνευση σε δύο μόνο ταμεία. Ευχαριστώ κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές. Ε, είναι καταπληκτική η παρουσίασή τους. Ε, συμφωνώ σχεδόν απολύτως με όλα αυτά που είπατε και είναι εξαιρετική βάση για να προχωρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. ο προπολογισμό θα πρέπει να ταιριάζει με το όραμά μα και να το συμπληρώνει. Και αυτό μπορεί να χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε τα πάντα από την αρχή. Δηλαδή αντί να ξεκινάμε από τις κατηγορίες, τον τίτλο, τίτλο σε 1, 2, 3 κτλ. και μετά να προσαρμόζουμε τον προπολογισμό σε αυτό, θα μπορούσαμε να επανασχεδιάσουμε ποιο είναι το όραμά μας, τι θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πηγαίνει πού όπως είπε η πρόεδρος Ρέντινγκ επανειλημμένα, έχει τονίσει ότι το νέο ε, μεγάλο ε, σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ένωση των Πολιτών. Αυτό είναι όραμα. Έρχεται ο προπολογισμό τώρα να ταιριάξει με το όραμα αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί σήμερα έχουμε το 1% δεν απατώμε για όλο αυτό το κλάδο ε, εσωτερικών δικαιοσύνης και ελευθερίας πώς θα είναι το νέο μεγάλο ε, όραμα μετά την εσωτερική αγορά τώρα η Ένωση των Πολιτών. Και με αυτό συνδέεται κάτι ακόμα. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης, σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη όταν προετοιμαζόμαστε για τις νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Γιατί καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι αποφασίσαμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και μετά το πρόγραμμα δράσης που απορρέει και αυτά. Σταματάμε εκεί. Και μπορεί ενδεχομένως οι πολιτικές να εφαρμόζουμε διάφορα πράγματα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό λαμβάνεται υπόψη, ούτε ξέρω σε ποιο βαθμό. Και θα ήθελα να μου κάνετε εδώ κάποιες διευκρινήσεις. Τώρα, άλλο θέμα σε ποιο βαθμό θα έχουμε ένα προπολογισμό που αυτή τη, τη φορά να μην ταιριάζει με το όραμά μας, αλλά με τις ιδιαίτερες ε, επιμέρους πολιτικές. Παράδειγμα, Frontex. Σήμερα ψηφίσαμε για τη Frontex και αποφασίσαμε ε, ο Frontex να έχει την εξουσία και τη δυνατότητα να ε, αγοράζει ή να νοικιάζει με leasing τον εξοπλισμό του. Αλλιώς, ακόμα και αν συζητάμε για ένα ελάχιστο χώρο ε, ή ελάχιστο όγκο ενεργητικών, είναι τεράστιο το κόστος και παραμένει τεράστιο. Από τώρα λοιπόν προγραμματίζουμε ε, τι θέλουμε για το Frontex στο μέλλον, ακόμα και για τα στοιχεία ενεργητικού, για την περιουσία τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον. Διότι όπως γνωρίζουμε η εντολή του θα επανεξεταστεί μετά από μία πέντα αιτία. Για τους οργανισμούς τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω. Ιδιαίτερα στη μετανάστευση δεν θα πρέπει να είναι αρμόδιες για τα ταμεία της μετανάστευσης. 13 οργανισμούς έχουμε του Frontex, τον Ιάσο τώρα και τέσσερα προγράμματα, τα μία μάλλον, που ε, ειδικεύονται Το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα θα πρέπει να παίζει ρόλο ο Frontex, να έχει λόγο για πώς δαπανώνται τα κονδύλια. Δεν είμαι βεβαίως ότι σήμερα έχει τέτοιο ρόλο. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει μάλλον. Ίσως αν έχει είναι έμεσος αυτός. Το ίδιο ισχύει για το ΙΑΣΟ. Ε, σήμερα έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες. Θα ήταν χρήσιμο κάπως να συμμετέχει και αυτό στη συμφωνία των κρατών μελών. Και τέλος, Συμφωνώ απολύτως με αυτά που ε, είπατε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κύριε Μανσελβίση, για προφανείς και αυτονόητους λόγους. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά θα πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της αλληλεγγύης μετά την έκτακτη ανάγκη. Παράδειγμα η Ελλάδα. Μπορεί σήμερα να μην είναι κατεπίγουσα η κατάσταση, αλλά σαφώς ε, μιλάμε ε, ακόμα και σήμερα για την αλληλεγγύη με την Ελλάδα, διότι οι επιπτώσεις τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να τα αντιμετωπίσει. Αυτά τα θέματα δεν έχουν εκλείψει. Ναι, για αυτά που είπατε για τις κατεπήγουσες ανάγκες, αλλά και περιστάσεις να το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Έχω πολλά να πω, αλλά έχω πάρει πάρα πολύ χρόνο και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσκεκλημένους μας, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ειλικρινής και απόψεις τους ήταν σαφέστατες, εναργέστατες. Κρίμα όμως που αφήσαμε αυτό το θέμα στο τελευταίο στην ημερήσια διάταξη και το συζητούμε τόσο λίγοι μεταξύ μας. Θα ήθελα να σας θέσω μία κοινή ερώτηση και απλούστατη, αλλά μετά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορώ να συνοψίσω σε μία μόνο ερώτηση. Σίγουρα θα πρέπει τα προγράμματά μας, τα ταμεία μας και τους πυλώνες μας να τα κάνουμε πιο φιλικά προς τα κράτη-μέλη και προς τους πολίτες, για να αντιληφθούν και οι χώρες και οι πολίτες τι κάνουμε εμείς εδώ. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αυτή η περίοδος προβλέπει κάποια κονδύλια που είναι φιλικά προς το χρήστη. Το, θε... το Ταμείο του, του Επαναπατρισμού είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ποιες είναι οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του άκουσα από την Επιτροπή ότι για το 2011 για την Ελλάδα δόθηκαν 25 εκατομμύρια από το Ταμείο Επιστροφής για να μπορέσει η Ελλάδα να επαναπατρίσει εθελοντές, ανθρώπους που ήθελαν και εθελώς να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι ξέρω, μόνο 800.000 θα χρησιμοποιήσει, 800.000 ευρώ θα χρησιμοποιήσει για την επιστροφή ε, των πάλι στον τον ελληνική κυβέρνηση. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση της εκταμίευσης αυτών των κονδυλίων από τα ταμεία ώστε όλα τα σχέδια που έχουμε και όλες τις στρατηγικές μας θα βοηθήσουν τελικά τα κράτη-μέλη και θα βελτιώσουν την απορρόφηση των κονδύλιων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βελτιωθεί ο βαθμός απορρόφησης και εκταμίευσης των κονδύλιων από τα ταμεία. Και τα ποσοστά που είπατε βέβαια και οι προπολογισμοί των ταμείων είναι σχετικά χαμηλοί και πενιχροί, αλλά παρόλα αυτά έχουμε κονδύλια που μένουν ανεκμετάλλευτα από τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα από τα κράτη που έχουν τις περισσότερες ανάγκες. Και παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούν στα έπακρα τα κονδύλια. Κυρία Σντάνοκα. Ευχαριστώ. Είμαι η τελευταία ομιλήτρια, mm. γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπαν η κυρία Κέλλαρ και ο κύριος Μπουσουτήλ για τα ταμεία. Άκουσα ότι υπάρχει πρόταση συγχώνευσης ε, των πέντε ταμείων σε δύο. Εγώ ήμουν κατά του κατακαιρματισμού, αλλά ήμουν ε, στη μειοψηφία. Εγώ είπα να μην ε, έχουμε ξεχωριστό ταμείο για την ισότητα των φύλων. Είπα να ενταχθεί αυτό το θέμα στην αρμοδιότητα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Η αντίθετη γνώμη όμως έλεγε ότι αν έχουμε πολύ γενικές αρμοδιότητες για τους οργανισμούς, τότε δεν θα καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα. Γι' αυτό έγινε ο καταμερισμός σε τέσσερα ταμεία ακριβώ για να μην αφήσουμε τίποτα στην άκρη. Τώρα εσείς ταχθήκατε μάλλον υπέρ μιας α, συγχώνευσης των ταμείων. Πώς όμως α, δικαιολογείτε την πρόταση για τη συγχώνευση. Πριν ξαναδώσω το λόγο στους δύο γενικούς διευθυντές, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Όπως βλέπετε, έχουμε μέλη στην Επιτροπή μας που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Και χαίρομαι για τα επιχειρήματα που μας δώσετε, γιατί μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στη συζήτηση στη ΣΟΥΡ. Και σίγουρα εδώ χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το σύνολο του επόμενου προϋπολογισμού, από το συνολικό κονδύλιο του κοινοτικού προϋπολογισμού και εκεί δίνουμε μάχη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιωθεί, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου και να βρούμε συμπληρωματικούς πόρους γιατί έχουμε και τη στρατηγική του 2020 και τις προτεραιότητες. Έχουμε και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχέδιο δράσης του προγράμματος Στοκχόλμης. Έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες, έχουμε όλο και περισσότερες κρίσεις που χρήζουν άμεσης και διεθνούς αντίδρασης και αντιμετώπισης, αλλά ταυτόχρονα υφιστάμεθα και την πίστη του Συμβουλίου που μας λέει να μειώσουμε τον προϋπολογισμό και όχι να τον αυξήσουμε. Εκεί ίσως θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μπορούσε να γίνει σύμμαχός μας στην προσπάθεια ενίσχυσης ή αύξηση του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για την κοινοτική προστιθέμενη αξία και αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο επιχείρημα ότι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχει προστιθέμενη αξία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και αντίστοιχα. Μιλήσατε για την ανάγκη ελαστικότητας και όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και καλό θα είναι αυτό το σύστημα με τους δύο πυλώνες να μην επιφορτιστεί από υπερβολική γραφειοκρατία και περίπλοκη χρηματοδότηση. Επίσης, θέλουμε η χρηματοδότηση να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα και να έχει στόχο την αποτελεσματικότητα. Επίσης, να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα συνεργειών και καλύτερου συντονισμού. Αναφέρθηκε η εξωτερική διάσταση. Όταν μιλούμε για την ασφάλεια, το θέμα της εξωτερικής διάστασης είναι πολύ σημαντικό. Και μιλούσαμε για τους τίτλους 3 και 4, για το ρόλο μας παγκοσμίως και του πόρου που έχουμε από την πολιτική γειτονίασης. Πώς πάει ο συντονισμό και τι είδου συνέργεια είναι δυνατή στα πλαίσια του επόμενου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί συζητήσαμε για τις έκτακτε ανάγκε και τις περιόδους κρίσης. Οπότε χρειάζεται κάποιο συντονισμό. Το θέμα του οράματος είναι πολύ σημαντικό. Αλλά στον επόμενο προπολογισμό θα έχουμε και τη στρατηγική του 2020. Και η ε, στρατηγική του 2020 έχει επικαλύψεις με όλες τις αναπτυξιακέ πολιτικές και με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Θα πρέπει να γίνει ένα είδος καλύτερου συντονισμού και συνδυασμού ώστε να αποφευθούν οι επικαλύψεις και να δοθεί έμφαση στη σύγκληση. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα να τα σχολιάσετε όλα αυτά. Ο κ. Μαλσερβίς, ευχαριστώ. Πρόεδρε, και για τις ερωτήσεις και για τα σχόλια. Ακόμα και αν έχουν προχωρήσει αυτά τα θέματα, ε, ε, διοργανώνουμε μια διάσκεψη στις 8 Απριλίου, ε, μια ακρόαση για να μπούμε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες από πολλά από αυτά τα θέματα. Όχι μόνο για το Κοινοβούλιο που είναι βέβαια και η σπονδυλική στήλη, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους δημοσιεύουμε και στην ιστοσελίδα μας ένα έντυπο για διαβούλευση μέχρι την Κυριακή που ολοκληρώνεται. Ε, συλλέγουμε στοιχεία και προτάσεις γι' αυτό προτείνω σε όσους ακόμα θέλουν να συμμετάσχουν να μην διστάσουν να το πράξουν. Και με πολύ μεγάλη χαρά ε, θα αφαιρώσουμε και ένα μικρό εργαστήριο σε αυτό το θέμα για να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το έχουμε ξαναπεί. Στα πλαίσια της διαδικασίας ε, που προωθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο, ε, η αφετηρία είναι αναθεώρηση του προπολογισμού, έτσι, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Το δεύτερο είναι η ανάγκη να ξέρουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι ανάγκες μας και σε περίοδους κρίσης, τι είναι προτεραιότητα και τι γίνεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλοι θα αποφασίσουν ε, το επίπεδο των πόρων και το ύψος των ποσών. Εδώ μπορεί να σας πω έτσι, μια προσωπική μου σκέψη ότι συχνά γίνεται λόγος για την προστιθέμενη αξία της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καμιά φορά ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το κόστος της μη Ευρώπης το λεγόμενο, ειδικά σε αυτούς τους τομείς είναι πολύ υψηλό το κόστος αν δεν κάνουμε μια σειρά πραγμάτων, έτσι, όχι μόνο πόσο κοστίζουν αυτά που κάνουμε. Ε, πάντως αυτό είναι το πλαίσιο όντως και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα είναι από τους βασικούς ε, πρωταγωνιστές. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν ε, ε, λόγο και εξουσία και ισχύ, αλλά και το Κοινοβούλιο επίσης. Δεν έθιξα κάποια ζητήματα βασικά γιατί είναι εκτός ε, των δικών μας αρμοδιοτήτων μέχρι στιγμής. Και ένα τελευταίο, σε ό,τι μας αφορά εμάς ε, συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο. Η συνθήκη τη Λισαβόνα ήρθε να επισφραγίσει και να ολοκληρώσει αυτό που στο παρελθόν λέγαμε κοινοτικοποίηση τη ε, δράση, ιδιαίτερα στην εσωτερική πολιτική. Τώρα έχουμε ε, ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία και συναπόφαση που είναι η συνήθις νομοθετική οδός αλλά και έχουμε και μεγαλύτερη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με τους γείτονές μας και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλούμε για το όραμα και τα εργαλεία ε, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την πολιτική ε, γειτονία, κύριε Άλβαρο. Σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής γειτονίας ασχολείται ακριβώς ήδη από τώρα με πολλά από αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω εάν ο στόχος εξυπηρετείται καλύτερα αν το βάλουμε σε ένα νέο τίτλο ή διαφορετικό. Αυτό είναι ένα θέμα επιλογής της μεθόδου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι περισσότερα από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να συνδέονται με ένα στόχο που εντάσσεται εκεί τις πολιτικές των εσωτερικών υποθέσεων. Και διάβασα και την έκθεση του κυρίου ε, Γκαρίγα, αλλά θα γίνει και μεγαλύτερη συζήτηση για την τελική δομή και αρχιτεκτονική. Αυτό μπορεί να είναι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει νόημα για ε, ε, περισσότερη ε, διαδραστικότητα και πιο περίπλοκη, έτσι πιο σοφιστική. Εμένα δεν με απασχολεί ε, τόσο πολύ αυτό, να δούμε πώς θα την προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Σε ό,τι αφορά αυτά που ρώτησε η κυρία Κέλλερ για τη ε, συνδιαχείριση. Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τις μεταρρυθμίσεις, γιατί στο κάτω-κάτω Ήδη υπάρχει κάποια συνδιαχείριση των ε, ταμείων, αλλά με ένα ε, παλαιομοδίτικο τρόπο όπου μοιράζουμε τους πόρους και μετά ελέγχουμε λίγο λογιστικά τους λογαριασμούς. Δεν είναι ακριβώς αυτό η συνυπευθυνότητα. Ε, πολλές φορές δεν ε, φαίνονται, δεν προβάλλονται σωστά γιατί δεν συνδέονται. Ορισμένα πράγματα γίνονται αλλά δεν το ξέρει κανείς. θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη διανομή καλύτερη προβολή και επέκταση. Γιατί νομίζω ότι εμείς θα πρέπει άμεσα να διαχειριζόμαστε λιγότερα, αλλά με μεταρρύθμιση με διαφορετικό περιβάλλον και περιεχόμενο. Για τις εξωτερικές δράσεις όχι, δεν συμφωνώ, δεν νομίζω. Γιατί η εξωτερική δράση θα πρέπει να διέπεται από τις ανάγκες που έχουμε για να υποστηρίξουμε κάποιες δραστηριότητες. Το θέμα τώρα στην εξωτερική δράση να έχουμε στη διαχείριση ε, η συνυπευθυνότητα όχι, χρειάζεται λιγότερο κατακαιρματισμό και μεγαλύτερο σχεδιασμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσουμε ε, σε κάποιου ειδικού και συγκεκριμένου στόχου. Τώρα, για το προπολογισμό τη εξωτερική δράση, πού πρέπει αυτό να ενταχθεί και αν τα θεματικά προγράμματα θα εξαφανιστούν. Κοιτάξτε, Κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει να εξαφανιστούν τα θεματικά ε, προγράμματα γιατί ε, η ανάπτυξη και η μετανάστευση είναι στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής και εκεί υπάρχουν πλεονεκτήματα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να καταργούμε προγράμματα, αλλά να συμπληρώνουμε την εργαλειοθήκη αυτή που λέμε με κάτι που δεν είναι αποκλειστικά ε, αφιερωμένο στην αναπτυξιακή πολιτική αλλά στις δικές μας ανάγκες γιατί εκεί προβάλλουμε τη δική μας πολιτική μετανάστευσης. Βεβαίως αυτά θα πρέπει να είναι ε, συμβατά, να μην φτιάχνουμε προγράμματα που να συγκρούονται μεταξύ τους, όχι. Αλλά η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική γιατί κυρίως τα μέσα που έχουμε είναι αναπτυξιακής κοπής να τα κρατήσουμε αυτά, αλλά να τα συμπληρώσουμε με κάτι άλλο που δεν είναι αμυγός αναπτυξιακό μέσο, αλλά μας βολεύει και μας για τη δική μας πολιτική και να είναι και κάπως συνεκτική η εξωτερική μας πολιτική. Για το σύστημα των δύο πυλώνων και ποιο είναι το πλεονέκτημα. Η πλούστευση, μεγάλο πλεονέκτημα. Αντί να έχουμε τέσσερις-πέντε νομικές βάσεις, να έχουμε μόνο δύο, είναι μεγάλη υπόθεση. κοινή διαχείριση αλλά με προσανατολισμό στους στόχους. Δηλαδή από μόνο το αυτό είναι τεράστια βοήθεια, απλούστευση και πλεονέκτημα. Έτσι θα έχουμε και καλύτερες συνέργειες και επιδράσεις. Στην πραγματική ζωή ο κόσμος δεν κοιτάει ε, <laughs> τα διάφορα ταμεία έτσι στην κάθε τη δομή τους δεν, ε, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Μιλάμε για στόχους που μπορούμε να ε, συνδυάσουμε. Στέγαση, εκμάθηση ξένων γλωσσών, βελτίωση ε, των δεξιοτήτων για οικονομικούς λόγους. Ε, μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη ελεγγύη σε συγκεκριμένες κοινότητες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με ενιαία μέσα και αν μπορεί κανείς να τα προγραμματίσει όλα αυτά από όλα τα μέσα, ενδεχομένω και από τα περιφερειακά ταμεία, γιατί όχι. Θα πρέπει να ανταλλάσσουμε εμπειρίες για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι τα ταμεία. Ε, ε αλλά τα ταμεία είναι μέσα για να εξυπηρετούν κάποιους στόχους που, που, που, που ζουν οι πολίτες καθημερινά και, και χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός και αλληλοσυμπλήρωση. Κύριε Μπουσουτήλ, για το απόλυτο ποσό ή το απόλυτο ποσοστό το 1%. Δεν είναι ε, αρκετό, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να σας πω ποσοστό. Τι να σας πω, θέλουμε 10%. Όχι, να συμφωνήσουμε πρώτα τους στόχους, να συμφωνήσουμε την προστιθέμενη αξία και μετά να αυξήσουμε το ποσό. Όραμα, προτεραιότητα και μέσα στη συνέχεια και τα λεφτά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πρόταση ε, για τις προτεραιότητες και τα ποσά εξορισμού είναι περισσότερα προφανώς αυτά που χρειαζόμαστε. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης λαμβάνεται πλήρως υπόψη, αλλά έχει και χρονικό ορίζοντα. Λίγη ε, με το πέρας των ε, τρέχουσών ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε, τι είναι πιθανό να κάνουμε και ποιες είναι αυξημένες ε, αρμοδιότητες, εξουσίες αλλά και ευρωπαϊκή διάσταση. Όχι μόνο το πρόγραμμα της Στοχόλμης, αλλά και λίγο πιο πέρα από το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Έρχομαι τώρα στους οργανισμούς. Frontex και EASO. Ε, συμφωνώ. Ε, καλό είναι που το Κοινοβούλιο έκανε την πρόταση για καλύτερο εξοπλισμό του Frontex το είχαμε σκεφτεί κι εμείς. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι αυτοί οι οργανισμοί τύπου Frontex και EASO να έχουν πιο συστηματικά μέσα στη διάθεσή τους για χάραξη πολιτικής. Έχουμε μια συστηματική κρίση η συστηματική ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να βοηθούμε τις χώρες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Ε, η κρίση σήμερα στην Ελλάδα, στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά ε, κάτι που να υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνει πιο αξιόπιστη τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Uh, um, λοιπόν, αυτά μπορούν να υποστηριχθούν από το ε, ΕΑΣΟ, την Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο. Και πάλι θέλουμε να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τελικά θα πρέπει να καταλαβαίνουν οι πολίτες τι κάνει η Ένωση, όχι αποσπασματικά. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι η υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιο άλλο οργανισμό, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι να φαίνεται η Ένωση. Και το θέμα των εκτάκτων καταστάσεων, των, των επιγουσών και και αυτό εκ των προτέρων να το έχουμε σχεδιάσει. Πώς να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια, να τα απορροφήσουν. Μα ήδη το πράττουμε. Από ό,τι φαίνεται, ε, όχι με εντελώ ικανοποιητικά αποτελέσματα, γιατί πολλά αυτά, από αυτά τα χρήματα υποαπορροφώνται, όχι μόνο στην Ελλάδα κατά τα άλλα, και αυτό δείχνει ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ακούμε τον κύριο Παπα-Νικόλα. Ε, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, είναι με καλή παρέα, γιατί και άλλοι δεν μπορούν να τα απορροφήσουν γιατί είναι υπερβολικά γραφειοκρατικοί όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, οι κατακαιρματισμένοι. Μπορώ να σας κάνω ένα κατάλογο ιδεών για το ε, πώς μπορεί κάποιος να κάνει ένα άκαμπτο εργαλείο εύκαμπτο πάντα στα πλαίσια του νόμου. Για την αξιολόγηση τώρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στην πλευρά της ασφάλειας ε, αξιολογήσαμε το πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο. Συλλέγουμε στοιχεία για κάποιες περιόδους. Είμαστε υποχρεωμένοι και πάλι με βάση την ομοθεσία αργότερα φέτος να υποβάλουμε την αξιολόγηση. Αυτό πάντα ως προθεσμία δεν ευθυγραμμίζεται με την πολιτική πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά θα πρέπει και εμείς κάπως να δικαιολογούμε, να ε, υποστηρίζουμε και αυτά που κάνουμε με ε, ένα σωστό ε, τρόπο αξιολόγησης. Αλλά δεν μπορεί η αξιολόγηση να έρχεται μετά τις προτάσεις. Πρώτα να γίνεται αξιολόγηση και μετά να διαμορφώνται οι προτάσεις. Είμαστε στη διάθεση όλων και του Κοινοβουλίου, αλλά μην ανησυχείτε τα εξετάζουμε. Και αυτά που λέμε δεν, δεν μας έρχονται ουρανοκατέβατα, βασίζονται σε στοιχεία. Εγώ θα προτιμούσα να έχω και παραπάνω στοιχεία, ο καθένας εργάζεται με αυτά που διαθέτει. Και ένα τελευταίο πρόεδρε. Σημαντικό αυτό που είπατε για το συντονισμό με άλλα ταμεία. Εγώ θα έλεγα εκτός ε, του, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών. Αυτό είναι θέμα όλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι θα πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε με έναν τρόπο πολύ πιο εγκάρσιο, ολοκληρωμένο. Πολλές φορές χανόμαστε στον κάθε το χαρακτήρα μας ε, και στα περιφερειακά ταμεία. Ε, κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσαμε να συνεργαζόμαστε με το Περιφερειακό Ταμείο, με το Κοινωνικό Ταμείο και ε, στις εξωτερικές σχέσεις η αποτελεσματικότητα και το τελικό προϊόν θα ήταν πολύ καλύτερο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αποσχιστικός ο καθένας στη γωνιά του. Συνεργασία. Με διάφορους τρόπους. Το έχω συζητήσει και με συναδέλφους από άλλους τομείς πολιτικής να ενισχυθεί αυτή η συμπληρωματικότητα, να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα προβλήματα με καλύτερη διάθεση. Βεβαίω αυτό είναι ένα εργοτάξιο, δεν έχει λήξει η υπόθεση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Λεμπάγ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω σε μια σειρά σχολείων, κυρίω αυτών του κυρίου Μπουσουτήλ για την ιδιότητα του πολίτη. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το μέλλον. Όπως είπατε κι εσείς, η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη σε αυτό το θέμα. Και άλλωστε είναι ένα είδος μη του Αριάδνης που το βρίσκουμε σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λαμβάνουμε και εμείς υπόψη φυσικά στις δικές μας αναλύσεις. Και το θέμα είναι επίσης πολύ σχηδές. Όταν λέω ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους, αυτό είναι η βάση πραγματικά της ιδιότητας του πολίτη. Πολύ συχνά έχουμε κάνει αξιόλογες ε, πράξεις, αξιόλογες δραστηριότητες, αλλά το αγνοούν, ε, το αγνοούν οι πολίτες. Δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα έχουν και άρα δεν μπορούν να τα ασκήσουν αποτελεσματικά. Πρώτα λοιπόν από όλα θα πρέπει να κάνουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους. Και στο θέμα της εφαρμογής των πολιτικών. Στη δικαιοσύνη πολλές πολιτικές έχουν άμεσο σύνδεσμο με την καθημερινότητα ε, των πολιτών από την στιγμή της γέννησης μέχρι τη στιγμή του θανάτου τους. Υπάρχουν θέματα διαζυγίων, κληρονομιών, θέματα ε, δικαιωμάτων ε, από, από γαμικές σχέσεις. Θέματα λοιπόν δικαιοσύνης έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα όταν κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και συμβολική αξία σε ό,τι αφορά την πολιτική μας για θέματα δικαιοσύνης. Και είπαμε ότι οι πολιτικές αυτές θέλουμε να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την εφαρμογή. Ε, μας ρωτήσατε να λαμβάνουμε υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Φυσικά. Και θα σας δώσω και ένα άλλο πολύ σημαντικό παράδειγμα που αφορά την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης προβλέπεται κάτι τέτοιο. Φυσικά θα είναι χρονοβόρα διαδικασία και θα καλύψει μάλλον το τελευταίο μόνο τμήμα του επόμενου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου και φυσικά θα είναι και κάτι που θα έχει το τίμημά του και θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στις συνέργειες και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα των συνεργειών και το μιλούμε για την ιδιότητα του πολίτη είναι ένα θέμα που σχετίζεται με τις πολιτικές τις δικές μας αλλά και με άλλες πολιτικές της Ένωσης. Έχει σχέση και με την εφαρμόγη του νόμου μας ενδιαφέρει ως Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης αλλά έχει σχέση και με την ενημέρωση. Έχουμε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, για παράδειγμα. Γιατί και η επικοινωνία είναι ένα απόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας. Και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες συνέργειες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί άριθμα παραδείγματα, όπου προσπαθούμε να συνεργαστούμε στενά με συναδέλφους άλλων διευθύνσεων. Μάλιστα πριν αναλάβω αυτή τη γενική διεύθυνση, είχα εμπειρία από σημαντικό έργο σε θέματα καινοτομία. Και εκεί, και για την καινοτομία, ε, συνδυάζουμε τόσε πολιτικές, Το είδαμε και στην ενιαία αγορά, το είδαμε και στο θέμα τη ιδιότητα του πολίτη. Είναι δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, ε, για μια γενική διεύθυνση να εργάζεται απομονωμένα. Καμία ενωσιακή πολιτική δεν νοείται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Υπάρχει αλληλεπίδραση και αυτό το θέμα των συνεργειών είναι πολύ σημαντικό. Και όλο και περισσότερο συμπεριλαμβάνεται στο έργο μας. Και στο θέμα του προπολογισμού για τα θέματα δικαιοσύνης και ιδιότητες του πολίτη, αυτό το θέμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο για τις ε, πραγματικά περιεκτικές ε, παρουσιάσεις που μας τροφοδότησαν με πολλά επιχειρήματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε διάφορα, οπότε σας εύχομαι όλους καλό Σαββατοκυριακό και ραντεβού και πάλι στις 11 και 12 Απριλίου. Καλό σας βράδυ.